Uh, Καλημέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Συνεδριάζουμε σήμερα ολόκληρη μέρα και αύριο ολόκληρη μέρα. Έχουμε πολύ μεγάλη μερίσια διάταξη, πολλά θέματα. Καλωσορίζω όλους σας και επίσης όσους μας ακούν πρωί-πρωί στο διαδίκτυο. Θα ήθελα όλους ιδιαίτερως να καλωσορίσω τον Όλεσόν, τον δανό μας Υπουργό της Προεδρίας ε, του Συμβουλίου. Στη συνέχεια θα σας το συστήσω εκτενέστερα. Ε, Δύο διαδικαστικά καταρχήν. Στα σχέδια ημερήσιας διάταξης που έχετε λάβει πρέπει να σας πω ότι χρειάστηκε να κάνουμε μερικές αλλαγές στη σειρά των θεμάτων για να μπορούν να είναι παρόντες και οι Ε, Το απόγευμα, αν δεν απατώμε, είναι η πρώτη αλλαγή. Ο κύριος Τσασκόφσκι από... θα 3.30. Ε, αλλάξαμε ε, το θέμα του με την... Ε, γνωμοδότηση της κυρίας Κόμη για την προστασία των φυσικών προσώπων είναι αύριο το απόγευμα στις 4. Αυτή είναι σημαντική αλλαγή, η πρώτη. Και επίσης έχουμε αλλάξει και τη γνωμοδότηση της κυρίας Βάισκερπερ για την χορύπανση από μηχανοκίνητα οχήματα, το θόρυβο ουσιαστικά. Λοιπόν, αύριο είναι οι ψηφοφορίες, θα σημίζω στις 9.30 Έχουμε πολλές σημαντικές ε, ψηφοφορίες για γνωμοδοτήσεις. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι θα είστε παρόντες. Ε, και οι συντονιστές συνεδριάζουν αύριο στις 5, στις 21 Ιουνίου, για να το γνωρίζετε αυτό. Για να πούμε τι συνέβη το πρώτο εξάμεινο. Just to let you know also that we have... Uh, Επίσης, Έχουμε και ένα νέο newsletter ενημερωτικό για τον Ιούνιο. Δίνω ένα προσωπικό αντίτυπο στον Υπουργό αφιερωμένο και αν πάτε και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας, του Κοινοβουλίου δηλαδή, ε, μπορείτε και να το κατεβάσετε με ζωντανές ε, συνδέσεις, live ε, σε όλα μας τα έγγραφα και άμα στείλετε τη ε, διεύθυνση σας ηλεκτρονική θα σας έρχεται όποτε εκδίδετε στο ηλεκτρονικό σας γραμματοκιβώτιο και θα είστε φίλος στο δίκτυο της Επιτροπής μας. Είμαι βέβαιος ότι θα σας εγγράψει το γραφείο σας για να παραμείνουμε σε επαφή και στη συνέχεια. Αυτά ήταν τα θέματα που είχα να σας πω. Υποθέτω εγκρίνεται η μερίσια διάταξη με αυτές τις αλλαγές, οπότε και προχωρούμε. Έχετε τα πρακτικά της συνεδρίασης 30 και 31 Μαΐου. Θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Λοιπόν, μετά από αυτή τη μακρά εισαγωγή και ζητώ συγγνώμη Υπουργέ, θα ήθελα και πάλι να σας καλωσορίσω θερμότατα είναι ο κύριος Όλε Σόν, υπουργό Εμπορίου και Ανάπτυξης της ε, Δανικής Κυβέρνησης και ήρθε να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα της Δανικής Προεδρίας και κάποιες σκέψεις από την άποψη της δικής μας Επιτροπής ήταν πάρα πολύ επιτυχής και πάρα πολύ αφοσιωμένη Προεδρία. Και ένα από τα σημαντικότερα ήταν η συνεχής του υποστήριξη και διαρκής. Όλα τα θέματά μας τα κάλυψε με τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικό. Τον έχω συναντήσει επανειλημμένα και εδώ στις Βρυξέλλες και στην Κοπεχάγη, όπου πήγα και ξέρω ότι πήγαν και άλλοι συνάδελφοι. Και επίσης και χάρη ε, στους συνεργάτες σας και τους δικούς μας εισηγητές καταφέραμε να προοδεύσουμε πάρα πολύ σε σημαντικά ζητήματα και αυτό είναι πολύ καλό και για την Επιτροπή μας και για την Ευρωπαϊκή Οικονομία και ε, αντανακλάται και από την προσοχή που του έχετε δώσει. Έβαλα και τη δανέζικη μου γραβάτα σήμερα για να σας τιμήσω ε, και θα συνεχίζω να τη φοράω. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η περίοδος. Α, η Μπερναντέτ Βερνιό έχει βάλει και το δανεικό ε, φουλάρι και είναι πάρα πολύ κομψή, Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε με χαρά, σας καλώ να μας ε, δώσετε τα συμπεράσματα, μοιραστείτε κάποιες σκέψεις και ενδεχομένω και κάποια θέματα στα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή και μετά τη λήξη της Προεδρίας. Παρακαλώ, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σήμερα για τον απολογισμό της Δανικής Προεδρίας. Ξέρετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να έρχεται κανείς στην αρχή παρά στο τέλος, γιατί σας ε, υποσχόμαστε πολλά και μετά πρέπει να γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων για να δούμε κατά πόσο μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε. Κάτι το οποίο δεν είναι ευνόητο τι κάναμε και τι καταφέραμε σε σχέση με τις αρχικές μας ε, υποσχέσεις. Καταρχήν, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορώ να υπογραμμίσω και να τονίσω ότι μπορέσαμε να προχωρήσουμε αρκετά, να προοδεύσουμε ως προς τον τομέα της υποστήριξης των καταναλωτών και είχαμε και επαφές με τον πρόεδρο, με τον κύριο Χάρμπορ, με εσάς. Ήταν ε, μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εκ του σύνεγγης. Μόλις αναλάβαμε την Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διένυε μια μεγάλη κρίση. Και ίσως αυτή ήταν και η μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε ότι δεν έχει παρέλθει η κρίση αυτό είναι ένα δεδομένο, αλλά προσπαθούμε να την διαχειριστούμε και να διαχειριστούμε τις προκλήσεις. Όπως σας είπα, προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της ε, προόδου και της ε, ολοκλήρωσης της αγοράς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βασιστούμε σε αυτούς τους δύο πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, ανάπτυξη. Στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού μίλησα για θέματα μεταφορών ιδιαίτερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπη διότι υπέβαλε την πράξη για την ενιαία αγορά με τις 12 νέες πρωτοβουλίες που μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Οι νέες πρωτοβουλίες προκηρύχθηκαν, είναι κομβική σημασία στο έγγραφό μας και το έγγραφο της Κομισιόν δηλαδή και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ως προς τρία θέματα. Καταρχήν τον κανονισμό ως προς την τυποποίηση. Ελπίζουμε λοιπόν να φτάσουμε σε συμφωνία και ως προς το venture capital και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία και σε τρία άλλα σημεία ως προς την ενιαία αγορά. Την οδηγία ως προς τα λογιστικά μας, το Connecting Europe και την επίλυση διαφορών online σε σχέση με τις διαφορές των καταναλωτών. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε ένα νέο σχέδιο ως προς την πράξη ενιαίας αγοράς στο εγγύς μέλλον. Ως προ την οδηγία για την τυποποίηση, σας είπα ότι στα πλαίσια της Προεδρίας φτάσαμε σε μία συμφωνία με τα άλλα θεσμικά όργανα, άρα μπορούμε να εγκρίνουμε αυτόν τον κανονισμό για την ε, τυποποίηση. Φτάσαμε σε έναν πολύ καλό ε, συμβιβασμό και έχουμε να κάνουμε με ένα πιο ευέλικτο σχήμα. Οι εγγύσεις θα είναι πιο θα είναι απλουστευμένες σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τα συνδικάτα θα μπορέσουν να, να συμμετέχουν στη διαδικασία τυποποίησης. Επίσης, η όλη διαδικασία θα είναι βραχύτερη, θα διαρκεί λιγότερο. Αυτό θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Και αυτό σημαίνει ότι οι τεχνολογίες και οι κανόνες θα είναι πιο προβλέψιμη. Οι επιχειρήσεις θα είναι πιο παραγωγικές και θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη το, τις εξαγωγές των επιχειρήσεων. Επίσης θα μπορούσαμε να δράσουμε οριζοντίως, δηλαδή πέρα από τα σύνορά μας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρμπορ και την κυρία Κομή, καθώς και όλους τους σκιώδεις για την εξαιρετική συνεργασία και την ε, ε, διάθεση συνεργασίας και εξέβρεση συμβιβασμών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια διαδικασία όπου η πρόσβαση στο κεφάλαιο ε, είναι αρκετά δύσκολη και πιστεύω ότι τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες, έτσι ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά. Έχουμε δύο κοινέ προτάσεις για καλύτερη απασχόληση και για να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Επίσης, στα πλαίσια της Προεδρίας θέλουμε να εξεύρουμε σύντομα μία συμφωνία συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν ένα απλό σχήμα ως προς τις διασυνοριακές συναλλαγές. Γιατί θεωρούμε ότι πολλές χώρες προβαίνουν σε επιγραμμικές αγορές, online δηλαδή, σε επίπεδο 40%. Πολλοί δεν θέλουν να προβαίνουν σε αγορές μέσω διαδικτύου. Επίσης, πολλοί αγοράζουν από εθνικά δίκτυα και όχι διεθνή. Θέλουμε να αλλάξουμε λοιπόν την προϋπάρχουσα σύσταση έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση και στην επίλυση διαφορών. Έτσι θα αυξήσουμε την ασφάλεια των επιγραμμικών συναλλαγών διατηρώντας το σύστημα όπως είχε λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Επίσης, το όλο σύστημα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει βασικές αρχές. Οι συνάδελφοι από την Κύπρο θα αναλάβουν αυτό το θέμα και είμαι σίγουρος ότι η Κυπριακή Προεδρία θα οδηγήσει σε μια συμφωνία με τη συνεργασία σας. Επίσης μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός του κανονισμού περί δημοσίων προμηθειών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις. Φτάσαμε σε μια συμφωνία, προχωρήσαμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας και όπως γνωρίζετε είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να έχουμε μια κοινή αγορά δημοσίων προμηθειών. Θελήσαμε να απλουστεύσουμε τη διαδικασία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τους διαγωνισμούς γενικότερα. Μιλήσαμε για τον πολλαπλό ρόλο των αγορών δημοσίων προμηθειών. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη το δίπτυχο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής και της οικονομικής. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα νέα αυτά κριτήρια. Επίσης, σε μία έκθεση προόδου στο Συμβούλιο, βρήκαμε τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο. Μιλάμε για την διαδικασία διαπραγμάτευσης στα πλαίσια Συμβουλίου Κομισιού και μας ενδιαφέρει να ξαναδούμε την πρόταση της Κομισιόν έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και την, την οδηγία και τον κανονισμό για τις ΔΕΚΟ. Ένα άλλο σημείο αφορά την κινητικότητα του πολίτη, δηλαδή την δυνατότητα να εργαστούμε πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια επεξεργαζόμαστε και την οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων. Και ήδη έχει επιτελεστεί πρόοδος. Έχουμε λοιπόν προχωρήσει ως προς τις οριζόντιες διατάξεις. Υπάρχει και το διαβοτήριο επαγγελματικών ευρωπαϊκών προσόντων, το οποίο έχει προωθηθεί. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και για την εργοδοσία και για τους εργαζομένους. Δεν είναι καθόλου εύκολο χρειαζόμαστε ένα υψηλό βαθμό λειτουργικό πλαίσιο και γνωρίζουμε ότι και η Κομισιόν μας βοήθησε αρκετά. Ας ελπίσουμε να επέλθει συμφωνία στο εγγύς μέλλον. Επίσης, μας απασχόλησε η οδηγία περιλογιστικών θέλουμε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων. Και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την ε, τήρηση λογιστικών βιβλίων. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι και το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συνεισφέρει στις εργασίες αυτές. Η Ιδανική Προεδρία Επίσης ασχολήθηκε με την ε, καλύτερη, μάλλον με ένα καλύτερο κανονιστικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο ως προς την ψηφιακή αγορά. Θα πρέπει να υπάρχει σε διαχείριση και υποστήριξη της ανάπτυξης. Από το 2012 η Ιδανική Προεδρία ενέκρινε συμπεράσματα σε σχέση με την ευφύη νομοθεσία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την ε, συμπερίληψη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει αρκετά. Όμως οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να λειτουργήσουν έμπρακτα. Θα πρέπει αυτός ο κανονισμός να είναι διαφανής και αποτελεσματικός έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Η Ιδανική Προεδρία εξάλλου κατά το άτυπο συμβούλιο της Κοπενχάγης του Φεβρουαρίου τόνισε τη, τα δεδομένα της ψηφιακής αγοράς και την ψηφιακή αγορά όπως πρέπει να εξελιχθεί. Αυτό αφορά και τις δημόσιες προμήθειες από το 2016 και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο θα πρέπει να αντικαταστήσει τις τιμολογήσεις επί χάρτου. Τα συμπεράσματα ενεκρίθησαν στις 30 Μαΐου. Εργαστήκαμε και ως προς τα μέσα που ήδη υπάρχουν για να απλουστεύσουμε τη διαδικασία και για τις δημόσιες προμήθειες και για την ψηφιακή αγορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε φτάσει σε πολιτική συμφωνία για, συμφωνία, για, έχουμε θέσει μια συμφωνία για έγκριση σε πρώτη ανάγνωση. Εδώ έχουμε τις βάσεις ενός συστήματος που θα λειτουργήσει πολύ καλά, θεωρούμε, και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι διότι οι δημόσιες αρχές επιτρέπουν τη διεύρυνση αυτού του συστήματος και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον κύριο Μπιέλαν, καθώς και του Σκιώδης για την καρποφόρα αυτή συνεργασία. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ και στο Roaming 3. Φτάσαμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι στα πλαίσια της ε, κινητής τηλεφωνίας μιλάμε και για ε, ανταλλαγή δεδομένων και βεβαίως η χρήση της τηλεφωνίας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια και με μια λογική τιμολόγηση. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο θέμα. Εμείς τονίσαμε αυτή την ε, πρόταση και προτεραιότητα και ελπίζουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, σε συμφωνία πριν από τη λήξη της Δανικής Προεδρίας, έτσι ώστε να τηρήσουμε τις προθεσμίες που μας επέβαλαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Το τελευταίο μεγάλο θέμα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι θα επιληθεί θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και για το ενιαίο δίπλωμα έβρεση τεχνίας, ιδιαίτερα ως προς τις ε, μεταφράσεις γύρω από αυτό το πακέτο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, δεν θα ήθελα να ε, επανέλθω σε επιμέρους ζητήματα φέρουμε μια μεγάλη ευθύνη Εάν θέλουμε να βγούμε από την οικονομική κρίση, θα πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα. Σας ευχαριστώ και με στη διάθεσή σας για απάντηση σε ερωτήσεις. Well, thank Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ανασκόπηση και ε, μας ενημερώνετε ε, για πολύ σημαντικά θέματα της Προεδρίας σας. Εφτά συνάδελφοι έχουν ζητήσει ε, το λόγο. Μέχρι τις 10 και 4 έχουμε... Οπότε θα ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις τρεις με τη σειρά που σήκωσαν τα χέρια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερη σειρά. θα ήθελα όμως να ζητήσουμε από την κυρία Σαλντεμόζε να κάνει την πρώτη ερώτηση μαζί με τον κύριο Γκάρτ είναι εξέχοντα μέλη από τη Δανία στην Επιτροπή μας αλλά ήταν και συγγήτρια για τα πρότυπα. Θα ήθελα να καλωσορίσω και ε, ε, την κυρία Τόμψον που ε, ήταν πρόεδρος της ομάδας εργασίας. Είστε λοιπόν εδώ όλη η ομάδα. Είναι η κυρία Κόρα Σαμπίτ που ζήσει το λόγο και ο κύριος Λόχεγκαρτ, αυτοί οι τρεις πρώτοι, μετά την κυρία Σάλτεμόζη είπαμε, και μετά θα σας πω ποιους άλλους έχω. Mrs. uh, Mrs. Um, uh, Rula, and Professor Correa de Campos, uh, and Mr. Copperati. Okay. Anybody else? Άλλος κανείς από αυτούς που ακούσατε. Όχι. Ωραία. Η κυρία Σάλντε Μόζε τότε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι, Υπουργέ, στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι ε, που έχω την ευκαιρία να το κάνω και σήμερα. Μας είπατε ότι είναι πάντα ενδιαφέρον να έρχεστε στην Επιτροπή μας και να βλέπετε αν περάσατε τις εξετάσεις μετά το τέλος της Προεδρίας. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Κατά εξοχήν η Ιδανική Προεδρία στην προστασία των καταναλωτών και στην εσωτερική αγορά έχει επιτελέσει πάρα πολύ σημαντικό έργο και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας. Ιδιαίτερα χαίρομαι για το σύστημα ΙΜΗ και την τυποποίηση που ήταν προτεραιότητα για σας. Ε, δεν ήταν απλό, αλλά ήταν καλό το αποτέλεσμα το ημίνη το σύστημα πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά. Και αυτό θα βοηθήσει στην πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τούτο λεχθένων θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το μέλλον της εσωτερικής αγοράς. Πότε θα έχουμε μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλύτερα και να μπορούμε να αξιοποιούμε το πλήρες δυναμικό σε δύο χρόνια, πέντε, δέκα ή μήπως ποτέ. Γιατί πάντα χρειάζεται βελτίωση το σύστημα. Αυτό ήταν το ένα. Και ένα ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Είπατε ότι είναι σημαντικό οι κανόνες που ορίζουμε να είναι αποτελεσματικοί αλλά και διαφανείς ε, Κάτι που με ανησυχεί συχνά και είναι κάτι που θα σας απασχολήσει και εσάς και στη συνέχεια στο Συμβούλιο είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε και χειριζόμαστε τους υφισταμένους κανόνες. Γιατί αφιερώνουμε πάρα πολύ καιρό στην νομοθεσία, αλλά αυτό που ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο είναι αυτά που ψηφίζουμε, νόμοι, οι κανόνες να τηρούνται και να εφαρμόζονται. Ε, και εκεί χωλαίνει η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ανομοιογενής η εφαρμογή στα κράτη-μέλη και αυτό είναι εις και των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Θα μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν πώς εργάζεστε στο Συμβούλιο και αν η Δανική Προεδρία, η Δανία μετά την Προεδρία θα εξακολουθεί να τα θέτει αυτά τα θέματα στο επίκεντρο. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως εξετάσεις τις περάσατε. Ευχαριστώ. Τρεις είπαμε να ομαδοποιούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχολικές εξετάσεις ήταν αυτά που είπατε, αλλά εντάξει. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω μόνο ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τώρα που όλοι μιλούν για την ανάπτυξη, εσείς ε, βάζετε την ανάπτυξη ε, ε, μέσω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Πολύ ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση στην περίοδο αυτή του εξαμήνου και παρακαλώ να παραμένει η εσωτερική αγορά στην μερίσια διάταξη γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθει η ανάπτυξη παρά τα όσα αντίθετα ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε για την ψηφιακή ατζέντα και για την εφαρμογή της οδηγίας ε, των ε, υπηρεσιών ε, και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ως και ό,τι γήτρια για το σύστημα προφόρησης για την εσωτερική αγορά, το ΙΜΗ, θέλω να σας πω ότι ήταν και εκεί πολύ καλή συνεργασία και στην πράξη για την ενιαία αγορά τη δεύτερη. Μια ερώτηση, απαντήσατε βέβαια ότι είστε πολύ προσιλωμένος ε, να ολοκληρωθεί το θέμα του κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγεί κανείς στην Ευρώπη, στους επιχειρηματίες και στον κόσμο, όταν είναι τόσο κρίσιμο θέμα και όλοι συμφωνούν ότι είναι προς όφελος όλων ε, και θα μειωθεί και το κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρές. Και οι πάντες συμφωνούν επί της ουσίας και έχουν συμφωνηθεί όλα διαπληκτίζονται τώρα οι κυβερνήσεις για τις έδρες, για τις γλώσσες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πολιτικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει το μήνυμα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έρθει ανάπτυξη. Και είναι πολύ σημαντικό να το προωθείτε αυτό μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίο σε αυτό το γύρο, άλλο εξέχον ε, μέλος της Επιτροπής μας από τη Δανία, ο κύριος Λόκεγκαρτ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ φυσικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τη συνεργασία που είχαμε ε, σε αυτό το εξάμεινο. Δεν θέλω να μιλήσω για εξετάσεις εγώ ή διαγωνισμούς, το έκαναν άλλοι πριν και φτάνει αλλά και ο ίδιος ο, ο πρόεδρος ε, ε, υπουργός ε, ανέφερε ότι ήταν δοκιμασία αυτή η περίοδος. Το έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας. Υπήρχαν δύσκολα θέματα προς πρόθεση και καλό ήταν που βοηθήσαμε και εμείς γιατί υπήρχε και μία απογοήτευση Και βοήθησε αυτή η στάση που δείξατε ρεαλιστική, το είπε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κοιτάξατε τι ήταν εφικτό και ε, φροντίσατε να ολοκληρώσετε τις προσπάθειες εκεί. Με ρεαλιστικούς στόχους. Τώρα που μιλούν όλοι για την ανάπτυξη και συμφωνούμε ότι πρέπει να έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και ε, με κάποιο χρονικό ορίζοντα και ε, με κάποιους ρυθμούς. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε και η κυρία Μόζε. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας δεν αισθανθήκατε ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις εξελίξεις, να βοηθήσουμε για να έρθει αυτή η ανάπτυξη. Γιατί εμείς ως βουλευτές δεν μπορούμε εύκολα να εξηγούμε στους πολίτες ε, αυτά τα θέματα. Μιλάμε για την κινητήρια δύναμη της οικονομίας που πρέπει να τη βοηθήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε μια νέα όθηση και νέα ορμή σε αυτή την προσπάθεια. Μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον η χρήση αυτής της λέξης «Προεδρία του Μαύρου Ψωμιού». Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια στο μέλλον για να διευρύνουμε το πεδίο μας. Το μαύρο ψωμί, ψωμί σίκαλης, κάνει πάρα πολύ καλό, δίνει ενέργεια. Όσο πιο πολύ ενέργεια έχουμε, τόσο πιο δραστήριοι είμαστε. Αυτό το νόημα είχε η χρήση της λέξης μαύρο ψωμί. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια ως προς την ε, Δανέζικη Προεδρία. Είναι αλήθεια ότι διανύουμε μία περίοδο που τα ταμεία του κράτους ας πούμε ότι δεν είναι γεμάτα. Είναι δύσκολο να αναπτύξουμε νέες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται μια πιο ελαστική στάση για να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη ενέργεια, για να μπορέσουμε να περάσουμε από τα λόγια στη δράση. Γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να εναρμονίσουμε τους κανόνες έτσι ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτό που ξέρουμε καλύτερα στην ε, παραγωγή προϊόντων που γνωρίζουμε να παράγουμε και θα μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε. Θέλουμε λοιπόν να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες ε, στην εσωτερική αγορά. Για μένα είναι σημαντικό αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δοθεί μια όθηση στην ε, αγορά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό. Αν καταφέρουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το δυναμικό, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιοποίηση αυτή προς όφελος της ανάπτυξης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε σε ποια πραγματικότητα ζούμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να <clears throat> αυξήσει την ε, ανταγωνιστικότητά της. Και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας παίζουν καθοριστικό ρόλο. Όλοι είδαν τη λεπτομερή εργασία της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη ε, δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο εγχώριο. Αυτό μας υποχρεώνει να δράσουμε γρήγορα. Χρειάζονται 36.000 ευρώ κατά μέσον όρο για τη δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. 2.000 ευρώ απαιτούνται στις Ηνωμένε Πολιτείες. 600 ευρώ στην Κίνα. Βλέπετε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα για τη δημιουργία προσκομμάτων σε ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσίτεχνίες. Ευτυχώς οι επικεφαλεί των κυβερνήσεων στο τελευταίο συμβούλιο μας ανέθεσαν το καθήκον της δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Διπλώματο Βρεσιτεχνίας κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας. Δουλεύουμε πραγματικά πάρα πολύ σκληρά. Αυτό είναι ένα σημείο πρωταρχικής σημασίας ε, για μας. Όλο και περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούν να υπάρξει ένα πακέτο ανάπτυξης που θα μπορούσαν και εκείνα να υποβάλουν στο Συμβούλιο. Και το βασικό σημείο εδώ είναι ένας, ε, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα βρεσιτεχνίας. Δεν κοστίζει τίποτα. Δεν, δεν καλούμεθα να βγάλουμε λεφτά από τα, χρήματα από τα ταμεία μας, απλά και μόνο να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Θα ζητήσουμε ε, διπλώματα ευρεσιτεχνία σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό θα δημιουργήσει θέσει εργασία. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κανένα απολύτω επιχείρημα υπέρ της διατήρησης αυτής της κατάστασης Το θέμα της έδρας του δικαστηρίου των διπλωμάτων <clears throat> δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για τη δημιουργία και τη διαχείριση του συστήματος. Ελπίζω λοιπόν ότι θα βρεθεί μια λύση. Δύο λόγια ακόμα. Θα να αναφερθώ στο μέλλον της εσωτερικής αγοράς. Βεβαίως το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί κομμάτι αυτής της εσωτερικής αγοράς είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προσελκύει και εταιρείε να έρθουν να εγκατασταθούν. Όταν έχουμε ένα ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ανταγωνιστικές τιμές. Εμείς θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση μετά από αυτή την Προεδρία. Το μέλλον μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επικεντρωθούμε σε τρία σημεία. Θέλουμε να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά, εφαρμόζοντας τους κανόνες οι οποίοι θα υιοθετούνται ταχαίως αλλά και ψηφιοποιώντα την εσωτερική αγορά. Μόλις υιοθετηθούν τα τρία αυτά σημεία ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να δώσουμε μία όθηση στην εσωτερική ε, αγορά. Αυτή ήταν η ημερησία μας διάταξη κατά τη διάρκεια της ε, ε Δανέζικης Προεδρίας και αυτό έχουμε πρόθεση να κάνουμε και στο μέλλον με μεγάλη χαρά θα έχουμε την υποστήριξή σας στο Συμβούλιο. Είναι κάτι που θα ευχαριστούσε ιδιαίτερα αυτή την Επιτροπή. Τα, οι επόμενοι τρεις ε, ομιλητές, κύριο Σφά, κύριο Βενιού και κύριο Ζούλα. Κύριο Σφά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ βεβαίως να συγχαρώ τον Υπουργό για τη Δανική Προεδρία δεν θέλω να κάνω εικασίε για τις επιτυχίες σας. Αν ήσασταν καλύτεροι στο Συμβούλιο Υπουργών ή στο ποδόσφαιρο, στο Euro, εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο Κόμη ε, για την εργασία της, για τον κανονισμό, για ε, την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Ξέρω ότι συνεργαστήκατε πάρα πολύ κι εσείς ε, για την εσωτερική αγορά και το πιστώνουμε πάρα πολύ αυτό στη Δανική Προεδρία. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ε, ήταν κάτι που θέλετε να αναδείξετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, ότι το έχετε ε, σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί ε, να έχει στο μυαλό του κατηγορίες, ε, να σκέφτεται με βάση κάποια επιτροπή ή ε, κάποιες πολιτικές. Αυτό εσείς το καταφέρατε, κάποιοι άλλοι όχι. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό είναι μια πάγια τακτική στο Κοινοβούλιο έρχονται εδώ υπουργοί που θέλουν να δείξουν σύγχρονοι και μοντέρνοι και λένε να τονωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο βεβαίως. Και όταν πάμε στη συγκεκριμένη νομοθεσία και ξέρουν εδώ οι συνάδελφοι να σας πούν πολλά. Ε, κάθονται και λένε ναι, ναι, εντάξει, θέλουμε ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά εδώ να μην αλλάξει η εθνική νομοθεσία και εκεί ακόμα λιγότερο. Και καταλαβαίνω και την... Ε, ε, διστακτικότητα, θέλετε, και την προθυμία της δανικής ε, προεδρίας ε, για ένα ενιαίο εμπορικό δίκαιο στην Ευρώπη, αλλά θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να προωθηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και ένα τελευταίο. Έχετε απολύτω δίκιο σε ό,τι αφορά την ευρεσιτεχνία. Ε, είναι η πιο φτηνή μορφή η ανάπτυξη. Αυτό που είπε και η κυρία Σάλτεμόζ, η εφαρμογή των ηλυμένων αποφάσεων θα πρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχεται αποτελεσματικά. Και θα μας άρεσε πολύ αν υποστηρίζατε και την ανακοίνωση του κυρίου Μπαρνιέ για την ανάπτυξη και την ε, τόνωση της. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερνιό, παρακαλώ. Merci, Monsieur le eh Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ τη Δανική Προεδρία ιδιαίτερα για το ρεαλισμό της, αλλά και για την προσοχή με την οποία μας άκουγε. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη να δουν συγκεκριμένα, όπως είπατε, αποτελέσματα. Για την κινητικότητα, επειδή εργάζομαι πάρα πολύ σε αυτό το θέμα ε, της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, είναι ένα από τα ε, μέσα που θα φέρουν την ανάπτυξη στην Ένωση και η κινητικότητα αυτή θα καταστεί ανάγκη, που ήδη καθίσταται ανάγκη για πολλούς νέους στην Ένωση. Μιλήσατε για ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο επαγγελματικών προσόντων ε, και δεξιοτήτων. Διαβατήριο είπατε. Αυτό είναι αντίστοιχο με την επαγγελματική κάρτα. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές σε σχέση με την επαγγελματική κάρτα που αναφέρει το σχέδιο οδηγίας. Και επίσης μιλήσατε για υψηλές προδιαγραφές, απολύτως απαραίτητες, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι και περισσότερη Ευρώπη, καλύτερη Ευρώπη, αλλά και με πολύ ισχυρή προστιθέμενη αξία. Εδώ σε αυτό το θέμα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ελπίδα ε, και εμπιστοσύνη ε, στους πολίτες που μπορεί να είναι καταναλωτές, πελάτες, εργαζόμενοι, ασθενείς και με τα εθνικά κοινοβούλια ε, συνεργαζόμαστε Χτες ήμουν ε, στη Γαλλία και εργάστηκα με τη Γερουσία και την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ε, και βεβαίως υπάρχει αρχή της επικουρικότητας, αλλά δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε θετική κινητικότητα για τους επαγγελματίες και το σύνολο των πολιτών, εάν δεν οδεύσουμε προοδευτικά προς ένα κοινό πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης. Εσείς αυτή την εναρμόνιση πώς την αξιολογείτε και αν έχετε και προθεσμίες για να φτάσουμε σε αυτή, θα με ενδιαφέρει πολύ όχι μένα και όλους να το μάθουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη Δανική Προεδρία για την καλή μας συνεργασία. Νομίζω ότι τώρα που είναι βαθιά οικονομική κρίση και αυξάνεται ο σκεπτικισμός απέναντι στην Ευρώπη, ε, με αξιώσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων όλο και περισσότερο για επικορικότητα. Εσείς με το ρεαλισμό σας ε, και την υφαλιότητα πετύχατε ορισμένα. Ε, για τις υπηρεσίες θα επανέλθω στα πρότυπα. Ε, προχωρήσατε χωρίς να φυγούν οι δέκο. Γιατί υπήρχαν μεγάλες επιφυλάξεις και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τη συμπερίληψη των οργανισμών κοινή ωφέλεια και των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια ε, ανοίξατε τις σημαντικές υπηρεσίες ε, για ε, τα πρότυπα χωρίς να θίξετε αυτό που θα ήταν πρόβλημα για τις 10. Ε, πολύ καλό αυτό. Επίσης, καλωσορίζω και το συμβιβασμό που βρέθηκε στο σύστημα ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά, IMI, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη προστασία των δεδομένων, γιατί στην αρχή στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή μας δεν συνέβαινε. Η Δανική Προεδρία πέτυχε περισσότερα σε συνεργασία μαζί μας ε, και δεν μπορώ παρά να το καλωσορίσω. Έχω όμως και μια παράκληση. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η ρύθμιση ε, των ελαφρών οχημάτων, δικύκλων, τρικύκλων, τέτρακύκλων. Εκεί έχουν κολλήσει λίγο τα πράγματα. Θα σας παρακαλούσα να το προωθήσετε μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να με επιτύχετε εσείς περισσότερα ε, από την επόμενη, την Κυπριακή Προεδρία, λόγω της πείρας σας και μόνο και θα σας παρακαλούσα να αξιοποιήσετε τις τελευταίες μέρες της Προεδρίας σας για να ρυθμίσετε και τους τύπους αυτών των οχημάτων, των ελαφρών επαναλαμβάνω, γιατί έτσι θα έχουμε λίγο περισσότερη εναρμόνιση στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και αυτό είναι απαραίτητο για τους καταναλωτές, άνδρες και γυναίκες. Well, we made considerable progress last Έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος ήδη από χτες το βράδυ και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Η Προεδρία μας γνωρίζει πολύ καλά και παρακολουθεί την κατάσταση που διανύει η Ευρώπη. Θα πρέπει να βρούμε μία να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση, σε μία σταθερότητα. γιατί όπως και για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου είχαμε επιλέξει μια ιδιαίτερη τακτική, πανευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, κατά της Γερμανίας. Και είδαμε να, που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η τακτική μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όμως για τις ερωτήσεις σας. Και θα πρέπει, να, κατανοήσουμε την, ε, το τι συμβαίνει στην αγορά. Θα πρέπει να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την εσωτερική αγορά Πραγματικά αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ. Έγινε μία αναφορά στην ψηφιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ασχοληθούμε με το θέμα της ψηφιακής αγοράς. Είναι ένας τομέας που θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία θα πρέπει να βελτιώσουμε την ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς και για τις επιχειρήσεις αλλά και προς όφελος των καταναλωτών. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές ε, στις δημόσιες αγορές ε, καθώς και πνευματική ιδιοκτησία, η ρύθμιση των διαφορών. Όλα αυτά αποτελούν ένα πακέτο που θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής αγοράς. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα όθηση στην εσωτερική αγορά. Ένα άλλο θέμα τώρα. Η οδηγία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Πράγματι, η Προεδρία μας θέλησε να εξασφαλίσει την πρόοδο αυτής της αναθεώρησης. Και πραγματικά προχωρήσαμε, δημιουργήσαμε μία ισχυρή βάση που οδήγησε στην απλοποίηση. Η ομάδα εργασία δούλεψε πάρα πολύ ως προς το σημείο αυτό. Ασχολήθηκε με το θέμα των διαβατηρίων και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι είναι ένα τομέα όπου υπάρχει διαφάνεια. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση για τι ρυθμισμένε αγορέ, για τα ρυθμισμένα επαγγέλματα θα επιθυμούσαμε να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδο σε αυτό το τομέα. Στην ε, ομάδα εργασία του Συμβουλίου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένες ε, διατάξεις. Οι εργασίε αυτέ θα συνεχιστούν υπό την Κυπριακή Προεδρία. Τα θέματα αυτά θίγησαν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου <clears throat> Ανταγωνιστικότητας στις 30 Μαΐου. Η Κυπριακή Προεδρία θα αναπτύξει τις δραστηριότητές της και θα κάνει μια προσπάθεια να προχωρήσει στο θέμα αυτό των επαγγελματικών προσόντων. Αυτά θα είχα να πω σε ό,τι αφορά το τελευταίο θέμα, κυρία Ρούλ. για την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα να αναφερθώ στην απογευματινή συνεδρίαση, αλλά νομίζω ότι ε, θα είναι καλύτερα να μιλήσει ο Υπουργός Μεταφορών, η τελευταία συνάντηση της Προεδρίας. Ελπίζω να ε, φτάσουμε σε ένα συμβασμό σε σχέση με τα ελαφρά οχήματα και νομίζω ότι κινούμαστε προς μία συμφωνία, φτάνουμε σε μία συμφωνία Τελευταίος γύρος και θα φτάσουμε, όπως είπα πριν, και σε κάποιο The Campos, Κοφράτη και Γκέπχαρτ. Νομίζω κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τονίσω την υποστήριξή μου προς την Προεδρία της Δανίας. Αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο από τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα μεταξύ Πορτογαλίας-Δανίας. Δεν συνδέονται το ένα με το άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα όσα επιτύχατε κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας που είναι πολύ σημαντικά τη συμμετοχή των συνδικάτων κατά τη διαδικασία τυποποίησης την υποστήριξη και ολοκλήρωση των αγορών ως προς τις δημόσιες προμήθειες και για τις ΔΕΚΟ, αυτό είναι ύψιστη της σημασίας για μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μέλλον των ΜΜΕ. Όλοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη κλειδί, όλοι μιλάνε για ΜΜΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο οικονομικός ιστός δεν απαρτίζεται μόνο από ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε, ιδιαίτερα τις ΔΕΚΟ. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις ΔΕΚΟ. Ε, ως προς το επιγραμμικό εμπόριο, νομίζω ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις ΜΜΕ και σας ε, ευχαριστώ και για το μεγάλο βήμα ως προς την περιαγωγή 3. Ξέρουμε ότι σε τέτοια θέματα υπάρχουν πολλοί, ε, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αντιτάσσονται στην ε, πρόοδο. Αντιμετωπίσατε και δυσκολίες ως προς το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Στη χώρα μου υπάρχουν προβλήματα από ένα μεγάλο όμιλο δικηγόρων οι οποίοι αντιτάσσονται σε αυτό το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνιών. Αντιτάσσονται, βρίσκονται πολύ κοντά σε μεγάλα επιχειρηματικά και πολιτικά κέντρα και μιλάνε για το υψηλό κόστος που εμπλέκεται σε, αυτά τα, σε αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα τεχνίας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να προωθηθεί και πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και το επιγραμμικό εμπόριο και να μιλάμε για ενιαία εμπορική σύμβαση, η οποία και αυτή θα πρέπει να προωθηθεί με τη σειρά της στο εγγύς μέλλον. Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς το μέλλον της ενίας αγοράς. Εσείς είπατε πολλά και συγκεκριμένα ως προς τα πεπραγμένα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ε, εμβαθύνουμε το ζήτημα. Ως προς τη σημασία της ενιαίας αγοράς κανείς δεν αμφιβάλλει. Και αυτό φαίνεται διότι εσείς κατά την προεδρία σας ασχοληθήκατε με συγκεκριμένα ζητήματα για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα όμως να σας πω ειλικρινά ότι αυτές οι δυνατότητες δεν θα αναπτυχθούν εάν δεν πλαισιώνονται θεσμικά. Μπορούμε να μιλήσουμε για εναρμόνιση σε αρκετούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ως προς την παραγωγική διαδικασία, τις εμπορικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα στα ισχύοντα πλαίσια των κανονισμών. Όμως υπάρχουν και θεσμικοί περιορισμοί. Όταν αντιμετωπίζουμε θέματα όπως τις μεγάλες οικονομικές δραστηριότητες ή και κοινωνικές, όπως για παράδειγμα το θέμα της ομοιομορφίας, της ενοποίησης των δημοσίων προμηθειών ή το σύστημα εκχωρήσεων, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ε, εκχώρηση κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διευρύνουμε την ενιαία αγορά. Έχω όμως την εντύπωση ότι πέρα από συγκεκριμένα όρια δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αν δεν αλλάξουν και οι συνθήκες. Πρόκειται για μία γνώμη σε σχέση με τις ε, διαβλεπόμενες εργασίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας με βάση την ε, εργασία σας αυτούς τους ε, προηγούμενους μήνες. Νομίζω ότι είναι πολύ προκλητική η ερώτηση και θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Η κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, και εγώ πιστεύω ότι στην εσωτερική αγορά Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη προεδρία. Και χαίρομαι που βλέπω ότι με τη δική σας ε, προεδρία δημιουργήθηκε μια προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής που φαίνεται, είναι αυτή. Και κρίμα που με το Σέγγεν μπήκε ένα τέτοιο αρνητικό πρόσημο στην προεδρία. Είναι μια πολιτική που έρχεται σε ε, κατάφορη σύγκρουση ε, με την ευρωπαϊκή πολιτική και στρέφεται προς τη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών. Και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε άλλους τομείς πολιτικής και στους τομείς που αναφέρατε εσείς. Αυτό με το γραφείο για τις ευρεσιτεχνίες, το δίκαιο για τις ευρεσιτεχνίε και κινδυνεύει να αναβαγίσει λόγω έδρας του δικαστηρίου. Μα αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα ε, το πιο σήμαντο, αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μας και όχι που θα εδρεύει το δικαστήριο. Στο μέλλον ε, τέτοια βήματα πρέπει να κάνουμε. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε κι εσείς γιατί περιμένω μια απάντηση για τη γενική συζήτηση στο Συμβούλιο. Πώς το βλέπει για ε, το περαιτέρω εξευρωπαϊσμό της εσωτερικής αγοράς. Ε, παράδειγμα με ένα ευρωπαϊκό ενοχικό δίκαιο ή δίκαιο συμβάσεων. Ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνεται ε, ένα εθελοντικό σύστημα. Αλλά μένα δεν μου αρέσει και είναι γνωστό αυτό γιατί δεν είναι ευρωπαϊκή απάντηση αλλά έρχεται να θεσπίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών δικαίων. Εκεί βλέπετε καμία δυνατότητα στο μέλλον ε, να προχωρήσει το Συμβούλιο. Γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι απόψεις. Αλλά εγώ θα προτιμούσα ένα πιο ευρωπαϊκό δρόμο όπως ε, κάναμε με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ιδιαίτερα ε, στον ψηφιακό χώρο να υπάρχει μεικτή εναρμόνιση. Εκεί ε, που υπάρχει δυνατότητα δηλαδή πλήρης εναρμόνιση και εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα έστω μια ελάχιστη εναρμόνιση. Αυτό θα ήταν ο πραγματικός ευρωπαϊκός δρόμος και όχι αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς βλέπετε στο Συμβούλιο ότι έχει μέλλον αυτός ο δρόμος να δοκιμήσει. Δίνω το λόγο στον Υπουργό για τις τελικές απαντήσεις και συμβουλές εν κατακλείδη. Ο Προεδρεύων. Νομίζω ότι θα ήταν πιο λογικό να πω καταρχήν ότι άκουσα με προσοχή τα επιχειρήματά σας και όλα όσα ελέγχθησαν ως προς το συμβατικό δίκαιο και τα θέματα που άπτονται του ενιαίου χώρου Σέγγεν. Κύριε Κοφεράτη, ως προς τις δύο ερωτήσεις σας για τις θεσμικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν. Βεβαίως, μιλάμε για θεσμικές αλλαγές οι οποίες πρέπει να επιτελεστούν. Βλέπουμε όμως πείρας ότι όταν αρχίζουν αυτές οι θεσμικές αλλαγές ε, έχουμε να κάνουμε με μία ευαίσθητη καθημερινότητα. Υπάρχουν πολλά θέματα επιτάπητος στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να αναζωογονήσει την εσωτερική αγορά και για να βρει λύσεις έμπρακτα έτσι ώστε ε, να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα ωραία μας λόγια. Πρόκειται για μία πραγματιστική προσέγγιση και αυτή μας κατήφθηνε κατά τις εργασίες της ε, Προεδρίας. Διαπραγματευτήκαμε πολλά και νομίζω ότι μπορούν να αρθούν πολλά προσκόμματα της εσωτερικής αγοράς. Πανηγυρίσαμε τα 20 χρόνια της εσωτερικής αγοράς και είδαμε έμπρακτα ότι θα πρέπει καταρχήν να τηρηθούν οι κανόνες που υπάρχουν ως προς τις δημόσιες προμήθειες. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη και νομίζω ότι για μια Ιταλική επιχείρηση δεν είναι εύκολο να έχει πρόσβαση σε μια Δανέζικη, αλλά ε, ηλεκτρονικά κανείς μπορεί να αναζητήσει τα δελτία έτσι ώστε να μπορέσει να υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Νομίζω ότι η ψηφιακή αγορά λειτουργεί πολύ καλύτερα με την οδηγία περί αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων μπορούμε να καταστήσουμε πιο ευέλικτη την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προβάλλουμε αυτή τη θέση. Κύριε Κάμπος, ο, υπάρχει ε, σύνδεσμος μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων Κανείς δεν το αρνείται αυτό, όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις τα καταφέρνουν καλύτερα από μόνες τους, ενώ οι ΜΜΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς, διότι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα. Στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ΜΜΕ είχαν δυσκολίες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να δράσουν αυτόνομα, ακόμα και χωρίς τις τράπεζες. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ΜΜΕ, διότι είναι πλέον καινοτόμες και δημιουργούν νέες θέσεις. Δεν πρόκειται για μια μανιχαϊστική προσέγγιση, δηλαδή ή μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ. Ως προς το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βεβαίως υπάρχουν μεγάλοι όμιλοι δικηγόρων, οι οποίοι επικρίνουν αυτό το σύστημα το ενιαίο σύστημα ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Το ίδιο κάνουν και οι μεταφραστές. Πρόκειται για καθαρά συντεχνιακά συμφέροντα. Είναι το δέντρο που κρύβει το δάσος. οι δικηγόροι κάνουν, βλέπουν ε, την ε, απλούστευση αυτού του πλαισίου και χάνουν εργασία. Αλλά θα έπρεπε να χαίρονται θα έπρεπε να χαίρονται γιατί επί της ουσίας υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα στην αγορά γιατί όταν πληρώνουμε έναν δικηγόρο δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη της αγοράς. Όταν όμως υπάρχει πρόσβαση στα, στο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μακροπρόθεσμα, οι δικηγόροι θα έχουν με περισσότερη εργασία, θα πρέπει να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγχουν τις εξαγωγές, τη δημιουργία εργασίας και ούτω καθεξής. Αλλά όλοι κοιτάν τα μικροσυντεχνιακά του συμφέροντα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι το δέντρο κρύβει το δάσος. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει και αυτό, αυτός ο μακροχρόνιος ορίζοντας, ο οποίος είναι προς όφελος όλων. Αυτή η, πρωτοβουλία κομβική σημασίας έχει μεγάλη σημασία διότι η αγορά θα μπορέσει να λειτουργεί με λιγότερες δαπάνες και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Προεδρίας και Επιτροπής σας έδειξε ότι οι προθέσεις μας είναι πολύ καλές, θέλουμε να προοδεύσει η εσωτερική αγορά, να γίνει πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική και είμαι πεπισμένος ότι και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα δρέψουν τους καρπούς αυτής της κατάστασης, αν και αναγνωρίζω ότι πολλά μέτρα δεν είναι δημοφιλή, βραχυπρόθεσμα. Αυτό το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι αν η κινητικότητα είναι μεγαλύτερη, εάν έχουμε ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τότε ε, θα υπάρξει και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Όλοι θα ευεργετηθούν. Ελπίζω να κρατήσετε να έχετε πολύ καλή ε, γνώμη για την Δανέζικη Προεδρία στο κατατήληξη των εργασιών μας. Well, um, Olison, thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. που ήρθε στο τέλος και στην αρχή της Δανέζικης Προεδρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδειξες πόσο καλά κατέχεις όλα αυτά τα θέματα. Φαντάζομαι ότι κατάλαβες από τις παρεμβάσεις το πόσο εκτιμήσαμε τις απαντήσεις που έδωσες. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και φανταζόμαστε ή μάλλον ελπίζουμε ότι θα έχεις λίγο χρόνο για να χαρίσει τον ήλιο στη Δανία. Εγώ θα πάω την ερχόμενη εβδομάδα, ελπίζω να διατηρηθεί η ηλιοφάνεια. Θα είμαστε σε επικοινωνία, σε θεωρώ φίλο της εσωτερικής αγοράς. Ελπίζω τον χρόνο που θα απομείνει στη θέση σου θα συνεχίσεις να βρίσκεσαι σε επαφή μαζί μας. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Okay, gentlemen, um, back to um, Επανερχόμαστε λοιπόν στην ημερησία μας ε, διάταξη. Έχουμε μία σειρά από θέματα για να συζητήσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ λίγο ησυχία. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε μια αναθεώρηση των τροπολογιών της γνωμοδότησης της κυρίας Βάισκοψ. Αυτή είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και αφορά την πρόταση κανονισμού για την οικοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η της, Δ. Βάις Κέρβερ, δεν ξέρω εάν κάποιος θα πάρει το λόγο. Η κυρία Ρούρεντ είναι εδώ. Εγώ είμαι σκέδος εισηγητής για την ομάδα μου. Θα κάνω αργότερα ορισμένα σχόλια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βάις Γκέρμπερ για να μας ενημερώσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να σας πω τι γίνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί παράλληλα με την ηχορύπανση ε, γίνεται η συζήτηση και στην αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή, ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, γι' αυτό καθυστέρησα, γιατί ο κύριος Ούσκι που είναι εισηγητής ε, συνόψης είναι και ο συνάδελφος Μέντες που θα έρθει φαντάζομαι εδώ. Ε, αγωνιστήκαμε πολύ με το χρονοδιάγραμμα για να προλάβουμε να ψηφίσουμε αυτή τη βδομάδα για να ε, μπορέσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος να έχει τη δική μας ε, γνωμοδότηση. Είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά τους, θέλανε να ψηφίσουν τον Ιούλιο, αλλά μετά από όλες αυτές τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και αφού το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει λάβει καθόλου θέση ούτε έχει προχωρήσει, ε, πρότεινε ο εισηγητής η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να αναβληθεί για το Σεπτέμβριο. Ε, ζήτησα και εγώ το λόγο και είπα ότι α, το είχαμε φανταστεί αυτό, αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε ε, προσαρμοστεί στο σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και πολύ νωρί είχαμε ανταλλαγέ με του σκιώδεις εισηγητές και εμείς θα ψηφίσουμε. Τι να κάνουμε, εμεί κάναμε τη δουλειά μας αυτή το πάνε Σεπτέμβριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές. Είναι πάρα πολύ επικοδομητική η ανταλλαγή που είχαμε. Δύο συνεδριάσεις με τους κοιόδης και μάλιστα πριν λήξει η προθεσμία για τις τροπολογίες και θεωρώ πάντα χρήσιμο να έχουμε ανταλλαγές ε, νωρίς, επιταχύνεται τη διαδικασία και μπορούμε να κάνουμε ε, συμβιβασμούς όχι τελευταία στιγμή. Δέκα είναι οι νέες επιπλέον τροπολογίες που κατατέθηκαν στην έκθεσή Σύμφωνο Συμφωνώ ε, σε όλες ε, τις τροπολογίες σχεδόν των συναδέλφων. Είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό και πρόθυμη. Τις υποστηρίζω και όλες έχουμε κάνει και κοινέ τροπολογίες με τους συναδέλφους Βέστφαλ και Χάρμπορ. Και στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών είπαμε που μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα τον άλλο. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ στα σημαντικότερα για μας θέματα από τη σκοπιά της ε, Επιτροπής ε, Προστασίας των Καταναλωτών. Θέλουμε περισσότερη ενημέρωση για τους καταναλωτές και περισσότερη διαφάνεια. Για μας γενικά σημαντικό. Υπάρχει ήδη σήμανση για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, για το θόρυβο που κάνουν τα ελαστικά που ήταν η έκθεση ΣΦΑΠ θυμάστε και ε, επίσης για την κατανάλωση καυσίμων. Εγώ τώρα θέλω αυτή η ενημέρωση για το θόρυβο να είναι κάτι που να βλέπουν οι καταναλωτές, να υπάρχει δική σήμανση δηλαδή. Για ποιο λόγο. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε διαφάνεια για τον τρόπο που λειτουργούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, ε, θα πρέπει με αυτή την προσπάθεια να ασκείται και πίεση στις βιομηχανίες για ε, καινοτομία. Και αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν πιέζουν και οι καταναλωτές να κάνουν λιγότερο θόρυβο τα αυτοκίνητα, γιατί... Ε, υπάρχουν ήδη ε, γειτονιές, ε, σε αστικές περιοχές που απαγορεύεται η κυκλοφορία, νυχτερινή κυκλοφορία των ε, προμηθευτών με φορτηγά εάν υπερβαίνουν ένα επίπεδο θορύβου ή εκπομπές. Λοιπόν, χρειάζεται αυτή η πληροφόρηση και για τους καταναλωτές και για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος τι λέει. γενικά είναι θετικά διακείμενη σε αυτή την πρόταση, αλλά προηγουμένως απαιτεί να υπάρξει μελέτη αντικτύπου. διαφωνώ και έκανα και τροπολογία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ζητάμε μελέτη αντικτύπου, αλλά αυτό δεν μπαίνει σε αυτόν τον κανονισμό γιατί δεν ταιριάζει ούτε νομοθετικά. Είναι μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια νομοθεσία να κάνει αυτή τη σήμανση. Εδώ είναι η αρχή και μόνο της συζήτηση τώρα. Για τα ηλεκτρικά οχήματα που είναι το δεύτερο σημείο σημαντικό και ενδιαφέρον για μας η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει εναρμόνιση των κανόνων για το θόρυβο των ηλεκτρικών ε, οχημάτων. Από πλευράς εσωτερικής αγοράς αυτό είναι ε, καλό, αλλά όταν έχουν χαμηλές ε, ταχύτητες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν κάνουν θόρυβο, σε μεγάλες ταχύτητες κάνουν. Και μάλιστα η Επιτροπή Περιβάλλοντος προτείνει οριακές τιμές που είναι πιο αυστηρές ε, για τα συνήθεια αυτοκίνητα. Για τους τυφλούς πεζούς όμως υπάρχει πρόβλημα με τα ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με το θόρυβο, το μη θόρυβο. Και εγώ ζήτησα ε, η ρύθμιση να μην αφορά πως δεν πρέπει να είναι ε, ο θόρυβος, αλλά πώς πρέπει να είναι ο θόρυβος. Δεν είναι διαδικασία Hughes σε αυτό το θέμα, αλλά η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος μας εμπιστεύεται. Ε, τώρα, για τα όρια του θορύβου, έχω κάνει κοινές τροπολογίες με την κυρία Βέστφαλ και τον κύριο Χάρμπορ και συμβιβαστικές, που αποκλίνω λίγο από την έκθεσή μου. Τα σημαντικότερα είναι για τους μακροπρόθεσμους στόχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μετά από διετία και μετά από πενταετία δύο βήματα. Εμεί έχουμε και ένα πιο μακροπρόθεσμο στόχο. Μια νέα πρόταση για τη διαφορά τη ταξινόμηση κατηγορίες των αυτοκινήτων και των οχημάτων γενικά. Η πρόταση της Κομισιόν παρελθούσα δεν ήταν καλή και νομίζω ότι είναι συναντικό αυτό. Χρειαζόμαστε πιο ρεαλιστικές τιμές. Εμείς είμαστε και πιο αυστηροί ε, αλλά και πιο ρεαλιστές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά. Οι τεχνολογίες που μπαίνουν για να μειώνουν το θόρυβο μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ή ακόμα και την ασφάλεια των οχημάτων ε, να επηρεάζουν. Γιατί αν υπάρχει αυτή η τεχνολογία που λέγεται encapsulation, που δεν ξέρω πώς το λένε στα γερμανικά για τους κινητήρες, να έχουν ένα περίβλημα, εν περιπτώσει, αυξάνονται και οι θερμοκρασίες. Και στα λεωφορεία διακυβεύεται και η ίδια η ασφάλεια ε, των ε, επιβατών. Γι' αυτό είναι πολύ καλή η τροπολογία της κυρίας Βέσφαλ, που στην αιτιολογική σκέψη ε, και σε αυτό αναφέρεται και τις οριακές τιμές για το θόρυβο. Και έχουμε και διάφορες φάσεις στον παραγωγικό κύκλο και προτείναμε και άλλες ε, Α, ήρθε ο συνάδελφος ε, Τόν Μάντερς ε, που προτείνει άλλες οριακές τιμές, ολόκληρη ταμπέλα, πίνακα. Αυτή είναι η μόνη τροπολογία που δεν έχω βάλει θετικό πρόσημο στον κατάλογο ψηφοφορίες για διάφορους λόγους θα το απέριπτα. Δεν έχει μακροπρόθεσμο στόχο, μόνο αυτή την πενταετία δεν έχει επιπλέον ας πούμε νέες τιμές και ε, μιλάει για διαφορετικούς κύκλους παραγωγής ε, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη το ότι άλλους κύκλους έχουν τα γιοταχή και άλλα τα φορτηγά και ένα ε, δεσιβέλ μόνο για τα οχήματα που είναι εκτός ε, δρόμου και πάλι δεν μου αρέσει. Είναι έξι διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ε, Volkswagen, Golf, Renault, Kangoo Electric. Είναι 68,4 δεσιμπέλ και εδώ προτείνονται 67 και κάτω. Μα αυτό δεν τα τηρούν ούτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πόσο μάλλον τα συμβατικά. Νομίζω ότι μέσα αυτές που αναφέρονται εδώ είναι υπερβολικά ε, ανεδαφικές και καθόλου ρεαλιστικές. Η πράσινοι λένε θα ψηφίσουν αποχή. Το δέχομαι αυτό. Σε αυτό. Και αν υπερψηφίσουν τελικά την έκθεσή μου θα χαρώ ιδιαίτερα. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις συζητητέ ε, για την πολύ ε, ευχάριστη συνεργασία όπως πάντα και ε, θα προσπαθήσω να υπερασπιστώ τις θέσεις μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως το έκανα και σήμερα το πρωί και ελπίζω να συνεισφέρουμε επικοδομητικά από πλευρά μα αυτή τη σημαντική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάσκεβε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, κύριο Μάντας. Μου φαίνεται ότι αναρώσατε. Χάσατε τη τριμερή συζήτηση βέβαια χθε. Παρακαλώ, κύριε Βέσφαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να ακρηγορήσω η κυρία Δόκτωρ Βάις Κέρμπερ τα είπε, ε, τα της συνεργασίας. Από την αρχή ήταν σαφές ότι σε πολλούς τομείς και ε, στη γνωμοδότηση και στην ανταλλαγή δείξαμε ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε, έχουμε την ίδια άποψη. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι προηγουμένως ακούσαμε επένους προς τη Δανική Προεδρία για την επικοδομητική και αποτελεσματική της στάση με εξαίρεση το Σέγγεν. Συμφωνώ απολύτω. Το πρόβλημα όμω είναι ότι χτε, για παράδειγμα, είχαμε διαπραγματεύσει τον τριμερή διάλογο ε, για ε, τα αυτοκίνητα ε, αυτά. Δεν είναι τόσο απρόσκοπτη η διαδικασία δεν έχουν ακόμα καταλήξει, δεν υπάρχει νομοδότηση. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας, ε, δώσαμε τα στοιχεία μας που είναι ε, σωστά και μεθοδικά. Αυτό φαίνεται και στις πολλές κοινέ τροπολογίες ε, που είχαμε. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να εγκριθεί και εδώ με μεγάλη πλειοψηφία. Η κυρία Βάις αναφέρθηκε προηγουμένως σε κάτι που με ενδιαφέρει και μένα πολύ. Ο θόρυβος των ελαστικών είναι ένα μόνο στοιχείο της αλήθειας. Το άλλο στοιχείο της αλήθειας που δεν αναφέρεται καθόλου είναι το οδόστρωμα. Ε, και αυτό είναι ένα θέμα των Δήμων και των κοινοτήτων. αυτό έχει δύο όψει στο νόμισμα, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, είναι και η άσφαλτος, ποιο είναι το οδόστρωμα που κυκλοφορεί. Γιατί έχει σημασία και αυτό. Σε όλη την Ευρώπη οι δρόμοι έτσι όπως αλφαστρώνονται συμβάλλουν στο θόρυβο και όχι στη μείωση του θορύβου. Ελπίζω πάντως να εγκρίνουμε την ε, γνωμοδότηση με μεγάλη πλειοψηφία και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Βαϊσπέργκερ και εγώ ήμασταν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να ακούσουμε αυτά που λένε και αυτοί εκεί. Και κατά την άποψή μου δεν έχει λήξει το θέμα. Εκεί πέρα συμφωνούν λιγότερο από ό,τι εμείς εδώ. Εγώ θα φροντίσω να περάσουν ορισμένες από τις τροπολογίες μου. Δεν βλέπω πολλές μεγάλες διαφορές ε, στις προτάσεις, ούτε τις δικές σας, Πρόεδρε. Και νομίζω αυτή είναι η άποψή μου. Και με, ε, με αναφέρουν οι εφημερίδες ως σκληρό υποστηρικτή της εσωτερικής αγοράς. Και εμένα με ενδιαφέρουν επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις δημιουργούν ευημερία και γενικότερα ανάπτυξη. Και η απασχόληση είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Είδα την νομοθεσία που κάναμε ε, υπό την ηγεσία του κυρίου Σφάπ για τα ελαστικά, αν θυμάστε, και γνωρίσαμε τεράστια πίεση από τα λόμπι της βιομηχανίας. Ότι αυτοί τα φτιάχνουν μόνοι τους τα ελαστικά και τα και μετά μας είπε η Μισελέν ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη και ε, ε, εμείς κανονίζουμε ε, τι κάνουμε, αλλά όταν έχουμε τέτοιες αυστηρές προδιαγραφές παγκοσμίως θα πρέπει να εισάγουμε ελαστικά από την Κίνα και από αλλού και θα χαθούν θέσεις απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για την πρόταση αυτή, αν μπορούμε να φροντίσουμε η ευρωπαϊκή αυτοκίνητο βιομηχανία να προχωρήσει με την καινοτομία της και να παράγει αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ε, σε σχέση με τους άλλους ε, κατασκευαστές αλλού θα είναι καλό και για την εικόνα της αγοράς της Ευρώπης και για την απασχόληση αλλά και για αυτούς που υποφέρουν από το θόρυβο που είναι 20 με 25% του πληθυσμού καθημερινά έρχεται αντιμέτωπο. Και δεν μιλάω για το φορολογούμενο που πληρώνει όλα αυτά τα ε, προστατευτικά που βάζουμε στους αυτοκινητοδρόμους, τα κράσπεδα και τα παραπετάσματα και όπως τα λένε όλα αυτά για να περιορίζεται όσο γίνεται ο κίνδυνος του αυτοκινητοδρόμου. Και ε, μπορεί να γίνει αυτό. Ε, το Δεκέμβριο ε, θα αρχίσει να ισχύει η νομοθεσία για τα ελαστικά και το 70% των αυτοκινήτων θα είναι κάτω των 66 δεσιμπέλ. Γιατί χρειάζεται διετία για τη βιομηχανία να προσαρμοστεί. Δεν 66, συγγνώμη, 67 δεσιμπέλ. 70 με 80% όλων των αυτοκινήτων ήδη είναι σε αυτό το επίπεδο. Γιατί θέλουμε μια διετία και μέσα σε πέντε χρόνια θα έχουμε φτάσει σε ένα ε, παραδεκτό επίπεδο και όλα αυτά γίνονται. Δεν θέλω να κάνω μια διάκριση με την πενταετία, αλλά ε, ο στόχος, ο τελικός είναι σημαντικός και μπορεί να επιτευχθεί βάσει των δικών μου προτάσεων αυτή την πρόταση που έχουμε εδώ τώρα στην Επιτροπή μας ε, τη θεωρώ χαλάρωση των ε, προδιαγραφών για το θόρυβο και το θεωρώ λυπηρό. Γιατί αποδυνάμωση και Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουμε την πίεση απέναντι στις βιομηχανίες. Θα πρέπει να φροντίσουμε για το μέλλον μας και για την οικονομία και για το περιβάλλον και για την ευημερία και την ε, ε, ευζοία των πολιτών μας. Με εξέπληξαν κάποιες δικές σας προτάσεις κύριε Πρόεδρε για τα φορτηγά. Όχι 80 δεσιμπέλ αλλά 82 δεσιμπέλ. Γιατί, πώς έτσι. Κάποιο λόγο θα έχει, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Κάτι άλλο που βρίσκω λιγότερο λογικό, ότι τα μίνιμπας πρέπει να είναι πιο αθόρυβα από ότι τα ταχύ. Και αυτό περίεργο, γιατί είναι μεγαλύτερα οχήματα κτλ. Την Πέμπτη θα ψηφίσουμε εδώ και καλά θα κάνουμε. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όμως ε, δεν έχουν πει τον τελικό τους λόγο και θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βάντες. Κύριε Συμφωνώ και συνεχίζω με αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Μάντερς. Θεωρώ ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για τις οριακές τιμές. Σε αντίθεση με τα ελαστικά, εμείς κάνουμε γνωμοδότηση μόνο και όχι οριστική θέση. Δεν είναι έκθεση. Η έκθεση είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Και η κυρία Βάις Γκέρμπερ το είπε και αυτή. Σε όλους τους τομείς όπου κατά την άποψή μου δεν είμαστε αρμόδιοι, θα πρέπει ε, να ψηφίσουμε εμείς αποχή. Δεν θα ψηφίσουμε την έκθεση σας, αλλά ούτε την εναλλακτική. Αποχή η ομάδα μου. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι κάνουμε προτάσεις για περισσότερη διαφάνεια, αυτό με τη σήμανση και το καλωσορίζω που δίνεται αυτή την όθηση, ακόμα και αν στην νομοθεσία δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει λίγο μια όθηση, μπας και ξεκινήσει. Και η εναρμόνιση για το θόρυβο των ηλεκτρικών οχημάτων είναι κάτι που συμφωνούμε οπωσδήποτε με τις προτιστάσεις σας και υποστηρίζω και αυτά που είπε η κυρία Βέστφαλ γιατί θεωρώ και ελπίζω να κάνει αυτή τη διαφορά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά επαναλαμβάνω δική μας ε, αρμοδιότητα δεν είναι να τα βάλουμε αυτά σε ιδεολογικές σκέψεις όχι στο διατακτικό. Uh, what a few comments. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Ναι, καταλαβαίνω ότι την είναι τελική ευθύνη, αλλά πιστεύω ότι η δική μας ευθύνη από την άποψη της εσωτερικής αγοράς είναι το να έχουμε μία σαφή και εφαρμόσιμη νομοθεσία. Πιστεύω ότι από τις ε, προτάσεις βελτιώσαμε το κείμενο. Πιστεύω ότι μερικές από αυτές αποτελούν μια πραγματική πρόκληση. Απαιτούν επενδύσεις. Είναι ένας πολύπλοκος τομέας, όπως ανέφεραν αρκετοί, γιατί υπάρχουν θέματα που αφορούν τα ελαστικά, αφορούν τους ίδιους τους κινητήρες των οχημάτων, Βεβαίως έχουμε δικαίωμα να έχουμε μία δική μας άποψη. Σε τελική ανάλυση όμως η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θα υποβάλει την πρόταση ανεξάρτητα από τη συνεργασία που θα έχουμε. Αλλά ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε μια μείωση του επίπεδου ε, της ε, ηχοστάθμης. Σε τελευταία ανάλυση αυτό που ζητάμε είναι οι κατασκευαστές να κάνουν επενδύσεις και να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες. Πιστεύω ότι υπάρχουν τομείς που θα μπορούσε να γίνει μια διαφορά. Να κοιτάξουμε μερικές από τις πτυχές της ενιαία αγοράς. Και από τη στιγμή που αυτή η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη και ήμουν εγώ υπεύθυνο για την ε, έγκριση της πρότασης, <clears throat> ένα από τα θέματα στα οποία εστιάσαμε την προσοχή μας, θα θυμούνται οι συνάδελφοι, είχε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης μικρών αλλά και μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Βεβαίω οι μικροί κατασκευαστές έχουν λιγότερους σπόρους, από την άλλη πλευρά συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους σε ό,τι αφορά την παραγωγή οχημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών. Αν ρίξετε μια ματιά στις τροπολογίες μου θα δείτε ότι ζήτησα της αναγνώριση της κατηγορία την οποία θα έχουν ε, πρόσβαση αναπηρικά αμαξίδια. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στα οχήματα για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αμαξίδια. Αυτή η τροποποίηση επηρεάζει πάρα πολύ τον ε, τομέα των οχημάτων και έχω την ε, εντύπωση ότι δεν εξετάσαμε παρκώς τι θα επιφέρει αυτό για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ευαίσθητοι για τα προαπαιτούμενα και αυτό ακριβώς κάνει η τροπολογία μου που ελπίζω να γίνει δεκτή. Ύστερα για αυτοκίνητα που παρουσιάζονται, ε, ε, ε, παράγονται σε περιορισμένο αριθμό. Θα έλεγα να υπάρχει ένας εκτενέστερος χρόνος προσαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το, το, το, το γενικότερο θόρυβο, τη γενικότερη πρόκληση θορύβου, αυτά τα αυτοκίνητα δεν ε, δημιουργούν πάρα πολύ θόρυβο. Εκείνα που δημιουργούν θόρυβο είναι τα εμπορικά και τα βαρέα οχήματα. Αυτά είναι ε, που επηρεάζουν περισσότερο τη ζωή των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά οχήματα, υπάρχει μια τεχνική τροπολογία Και πάλι ως θεματοφύλακες της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς ενημερωθήκαμε ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν ευθυγραμμισμένη με τις προτάσεις από την Ηνωμένα και την Γενέβη ως προς το συγκεκριμένο αυτό τομέα, όταν ετέθη το θέμα των ελαφραίων οχημάτων. Κάτι βεβαίω το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω εξέταση. Αυτό όμω δεν τα αφορούσε ως κατηγορία. Η τροπολογία μου λοιπόν η 23 που ελπίζω να υιοθετηθεί είναι μια τεχνική τροπολογία που επιλαμβάνεται αυτού του θέματο. Λέει ότι δεν η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει την ε, τροπολογία ε, την, ε, τον κανονισμό των Ηνωμένων και τη Γενέβη. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την στενή συνεργασία. Όπως είδατε, ε, έχω υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες, ελπίζω να εγκριθούν αύριο και μετά θα, η κυρία Βάσκε θα έχει το καθήκον να υπερασπιστεί την άποψή, την άποψή μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Όχι. Ωραία. Έχουμε χρόνο για να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Θέλετε να πείτε κάτι. Ζητάω συγγνώμη που δεν σας καλωσόρισα νωρίτερα. Και θα ήθελα επίσης ε, να σας ευχαριστήσω για το ρόλο που διαδραματίσατε στην τριμερή συζήτηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, μέσα στα προαπαιτούμενα για τη δουλειά μας είναι να είμαστε διακριτικοί. Δύο παρατηρήσεις σχετικά με τα όσα είπατε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία συνοχή στον τομέα αυτό και σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία της Γενέβης. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Αρχικά θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι απλό το έγγραφο. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλό το να προσπαθήσει κανείς να επιγραμμίσει την κοινωτική νομοθεσία με την νομοθεσία της Γενέβης. Αλλά καταρχάς πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση και αν θέλετε να επιστήσετε την προσοχή σε τομείς που δεν υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να υπάρχει μια διεθνής εναρμόνιση σχετικά με το θέμα της ε, ηχοστάθμη. Το, το ίδιο αφορά και τις βασικές αρχές ε, για την εξομοθεσία στη 2046. Αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα αναφερθούμε σε στοιχεία που αφορούν την ηχοστάθμη. Αν δεν είναι σαφές το κείμενο, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε το ε, ε, πλαίσιο, γιατί θέλουμε το σύστημα να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, είμαστε στη διάθεσή σας να το αναθεωρήσουμε, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίο. Αυτός ο φόρος θα πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητο, ε, ε θεωρείται απαραίτητος μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσει να γίνει αυτό και να ε, ληφθούν υπόψη και οι δύο αυτές πτυχές. Κύριε Βάσκα, Θέλετε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και βεβαίω. η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, θα πάω με χαρά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, να υπερασπιστώ την γνωμοδότησή μας και ο, ο εισηγητής ε, Όσκι ε, συμφωνεί να λάβουμε υπόψη και τα όσα προτείνουμε. Ε, είμαστε σε μόνιμη επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές εμείς εστιάζουμε στην επισήμαση και στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία. Να πω κάτι μόνο σχολιάζοντας τα όσα είπαν οι σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Βέσφαλ μίλησε για το δόστρωμα. Προφανώς θα πρέπει πάντα να υπάρχει η ίδια ποιότητα και να εφαρμόζουμε και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα παντού και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το συζητούν πολύ εντατικά και ο κύριος Ταταρέλα του ΕΦΤΑ και ο κύριος ε, Ούσκι. Ε, ε, υπάρχει και ιδέα που συζητείται για την ταξινόμηση των διαφόρων οδοστρωμάτων και να βελτιωθούν και οι ασφαλτοστρώσεις. Αυτό βέβαια μπορούμε να το ζητούμε, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι να το κάνουμε πολύ συχνά αυτό είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και έχουν προβλήματα και οι χώρες οικονομικά και οι δήμικοι κοινότητε. κοινότητες, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή σε αυτό. Εμείς μιλούμε για τα αυτοκίνητα που είναι κινούμενα προφανώς και κυκλοφορούν παντού. Ε, για το συνάδελφο Μάντερς, πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τις οριακές τιμές, το αποτέλεσμα θέλουμε το ίδιο. Μείωση του θορύβου, ανεξάρτητα από το αν προτείνουμε διαφορετικές τιμέ. και πίεση ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία για καινοτομία. Ε, παρένθεση. Ε, η δική μου πρόταση για τις οριακές τιμές είναι πιο φιλόδοξη από εκείνη του σκιώδους εισηγητή ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, κρίνει παρένθεση. Και οι συνάδελφοι Χάρμπορ και Βέστφαλ το βλέπουν όπως και εγώ συνολικά. Και δεν μπορούμε να πούμε έτσι ομά ότι εντάξει η βιομηχανία γενικότερα να κάνει περισσότερα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πιέσουμε εμείς, γιατί αν είναι υπερβολικά αυστηρές οι τιμές, τότε ενδεχομένως μπορεί να ε, οδηγήσει σε αύξηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και έχουμε και το πρόβλημα της ασφάλειας των οχημάτων. Ας πούμε, στα ελαστικά, εάν κάνουμε νέες ε, εγκοπές για να είναι πιο αθόρυβα. Δεν ξέρουμε τι πρόσδεση θα έχει στο οδόστρωμα μετά το κράτημα του ε, ελαστικού. Ε, και θα πρέπει ε, να έχουμε ένα μέσο όρο στις οριακές τιμές και όταν δεν υπάρχει αυτός ο μέσος όρος να πληρώνουν πρόστιμα οι κατασκευαστές. Και ο, κανονισμός αυτός από πλευράς κυρώσεων είναι πολύ πιο ε, αυστηρός γιατί ένα αυτοκίνητο που δεν καλύπτει ε, τις οριακές τιμές τότε ε, ε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο ολόκληρο. Δηλαδή δεν θα εγκριθούν αυτά τα οχήματα και μπορεί να είναι και το 70% των οχημάτων αυτό, ε, των ηλεκτροκίνητων. Δεν ξέρω, το λέω ίσως πολύ προσεκτικά, αλλά σε μια χώρα που παράγει αυτοκίνητα το βλέπει κανείς διαφορετικά από ότι σε μια χώρα όπως την ε, Ολλανδία που πρέπει να υφίσταται το θόρυβο. Αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Ε, θα υπερασπιστώ και πάλι την πρότασή μου, αλλά έχει δίκιο και η κυρία Ρούλε. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτά τα πράγματα. Αλλά και αν είναι πολύ ε, χαμηλές οι οριακές τιμές και αυστηρά τα όρια, θα αυξηθούν οι τιμές. Δηλαδή, ε, του αυτοκινήτου για τους καταναλωτές. Ε, και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά οι πράσινοι είπαν ότι θα ψηφίσουν αποχή γι' αυτό. Θα χαιρόμουν πάντω να υπερψήφιζαν την τελική γνωμοδότηση και για την πρόταση του παραρτήματος 3 τουλάχιστον να μπορούν να συμφωνήσουν σε μεγάλο βαθμό. Για τον συνάδελφο Χάρμπορ να πω ότι στην τροπολογία του 23 αλλά και τις άλλες έχω βάλει θετικό πρόσημο στον κατάλογο ψηφοφορίας, δηλαδή υπερψήφιση. Και ιδιαίτερα αυτό που προτείνεται για αυτοκίνητα που μεταφέρουν ανθρώπους με αναπηρίες. Και είναι σημαντικές οι προτάσεις σας, τις οποίες ε, ενστερνίζομαι. Αυτά ε, και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις για την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι δείχνει και πάλι η έκθεση ότι εάν ε, από νωρίς ανασκουμποθούμε όλοι μαζί και βοηθήσουμε, ίσως να συμφωνήσει εδώ και ο κύριος Μάντερς, μπορούμε να καταλήξουμε ε, σε κάτι και να κινήσουμε τα πράγματα σε αντίθεση με άλλες επιτροπές. Και αυτό ήταν κάτι που με ικανοποίησε και σε αυτή την νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο το πρωί. Ε, ελπίζω και σήμερα αργότερα για άλλα θέματα. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί λοιπόν τη γνωμοδότησή σας. Θα αρχίσει η ψηφοφορία στις 9.30 και μετά θα πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ψηφίσουν στις 10 ε, Ιουλίου. Υποθέτω ότι καθυστερούν κάπως την ψηφοφορία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ωραία, τελειώσαμε ε, με αυτό το θέμα. Είμαστε στην ώρα μας και περνάμε στο επόμενο θέμα, μία γνωμοδότηση και πάλι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο κύριος ε, Μπέκερ είναι η συγητής. Η κυρία ε, Χάνς Λίκ δεν είναι παρούσα, άρα ο κύριος Φαμπ θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ε, βλέπω ότι η κυρία Πέρες είναι εδώ, ο κύριος Χατζη η κυρία Ρούλ, η κυρία Μακλάρκιν είναι παρούσα, άρα έχουμε σχεδόν απαρτία. Ε, ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν είναι εδώ. Ας δούμε τι θα μας πει ο κύριος Σβάμπ, ο οποίος θα παρουσιάσει τη θέση της κυρίας Χάνσλικ και θα ακούσουμε και τους Κιώδης. Θα ψηφίσουμε αύριο. Κύριε Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ομολογώ ότι ε, αυτό που είπατε τώρα το acting report, ε, ε, ο ασκών καθήκοντα εισηγητού με τιμά και το ασθενίζουμε. Απλώς το μόνο που μπορώ να σας πω σήμερα είναι αυτά που μου έδωσε η κυρία Χάνσλικ για να σας παρουσιάσω. Δεν έχω αναλάβει την έκθεση. Ε, είναι συντάκτρια γνωμοδότησής μας η κυρία Χάνσλικ και δυστυχώς σήμερα κολλείται. έχει άλλη ενηλμένη υποχρέωση. Κυρίες και κύριοι, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που εγγράφονται στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα της Κομισιόν έχουν τεράστιες δυνατότητες να βοηθήσουν για την οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις απασχόλησης στην εσωτερική αγορά. Αλλά χρειάζονται βεβαίως ένα θετικό επιχειρηματικό κλίμα για να μπορούν να εργάζονται και να ε, ασκούν αυτή τη δραστηριότητα με όφελος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αν στο δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να ενισχύσουμε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες και να τις λάβουμε υπόψη γιατί έχουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως το δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, για την ανάθεση χρειαζόμαστε ε, ίσους όρους για να μην έχουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό θα πρέπει ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη ε, στη γνωμοδότηση αυτή ότι χρειάζονται ειδικέ προδιαγραφές για ειδικέ συμβάσεις με μία κατηγορία επιχειρήσεων που τα ε, αγγλικά λέει τις advantage persons που δηλαδή απασχολούν ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και θα πρέπει να ενταχθούν και αυτές οι απαιτήσει ε, όταν πρόκειται για ανάθεση συμβάσεων. Και η κυρία και ενδιαφέρεται να αναπτυχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, αλλά με μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική που να περιλαμβάνει όλη την Ευρώπη και να δίνει και δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας ε, και πρόσβασης τέτοιων επιχειρήσεων. Η γνωμοδότηση της κυρίας Χάνσλικ επίσης προτείνει η σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων να αναγνωριστεί. Γιατί γίνεται λόγος για κατανόηση ειδικών καταναλωτών ε, και ειδικών ε, αναγκών, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Το λέω γιατί με ακούει η συνάδελφος Ριγκόγεν είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές όπως αναφέρονται. Vulnerable consumers. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν τις δυνατότητες να συνεισφέρουν να διατηρήσουμε σε όλη την Ευρώπη ε, κοινωνίες των πολιτών ενεργές δραστήριες για να απαντήσουν στις δυσκολίες της οικονομίας και να βοηθήσουν για μια ανάπτυξη ε, ευρύτερη που να συμπεριλαμβάνει, να εντάσσει ε, όλους τους τομείς κοινωνίας. Inclusive growth το λένε αυτό στα αγγλικά η φιλελεύθερη μας υποστηρίζει, η δική σας ομάδα επίσης πρόεδρε, συντηρητική, με, αντίθεση, με εξαίρεση την πρώτη τροπολογία που πρόκειται για τις μικροπιστώσεις εκεί. θα τα ακούσουμε και στη συζήτηση και ελπίζω ως υπηρεσιακός ε, συντάκτης νομοδότησης να ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες σας. Ναι, πράγματι, ανταποκριθήκατε. Θα ε, συνοψίσετε βεβαίως ως ασκόν καθήκοντα εισηγήτη. Αρχίσουμε με τους ε, ε, ε Πέρες, ε, Χατζημαρκάκης, Μακλάρκιν, Ρούλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν κυρία Πέρες. Σας ευχαριστώ γιατί αναφερθήκατε στους ευάλωτους καταναλωτές γιατί πιστεύω ότι ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Χάνσλικ γιατί ήταν ιδιαίτερα ευέλικτη και δέχτηκε αρκετές από τις ε, τροπολογίες που υποβάλαμε. Φτάσαμε σε έξι τροπολογίες συμβιβασμού που είναι ύψης της σημασίας για μας. Στην παράγραφο 1 μιλάμε για ένα αριθμιστικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει την ιδιαιτερότητα και την προαγάγει, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιάζοντα χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να προσαρμοστούμε καλύτερα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και μιλάμε για βιωσιμότητα. Στην παράγραφο 2 μιλάμε για την ανάγκη να επιμείνουμε έτσι ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη ως στόχο έχω την ικανοποίηση των ε, κοινωνικών αναγκαιοτήτων ή γενικού συμφέροντος λαμβάνοντας υπόψη ε, την ε, σωστή συμπεριφορά το, τη σωστή συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη. Στην παράγραφο 4 μιλάμε για μια δική μας τροπολογία έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ενεργός κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη τη μία κοινωνία μη αποκλεισμών και την αλληλεγγύη και την ίση πρόσβαση μεταξύ ανδρών και γυναικών και την συμπερίληψη ε, πολιτών με ιδιαίτερες ανάγκες και την συμφιλίωση της ιδιωτικής, οικογενειακής και ε, επαγγελματική ζωή. Στην παράγραφο 6 μιλάμε για ένα νέο καθεστώς για τις κοινωνικές υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, έτσι ώστε οι τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνε για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων να προωθήσουν την κοινωνική ε, συμμετοχή και στην τελευταία παράγραφο μιλάμε για την σημασία άρσης προσκομάτων έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική δραστηριότητα και οι κοινωνικές προδιαγραφές οι οποίες ε, μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς κρίσης. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε στην ε, διευκόλυνση και την μείωση του διοικητικού φόρτου. Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι με βάση τις ε, τροπολογίες μας που δεχτήκατε θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τις ε, περισσότερες τροπολογίες που έχουν προβληθεί και υποβληθεί. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χάσλικ, έστω και την απουσία της, ε, και να την ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία συμπεριέλαβε όλους τους συζητητές, κατέθεσε ένα πολύ καλό κείμενο, αφετηρία, ισορροπημένο, ε, συμπεριέλαβε όλες τις ανησυχίες. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να είναι ε, σημαντικές για την καινοτομία, για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν δημιουργούν μόνο θέσεις απασχόλησης, αλλά είναι σημαντικές και για την κοινωνική συνοχή σε μια κοινωνία. Και αν δει κανεί ε, τις εξελίξεις στην Ευρώπη, διαπιστώνει ότι αυτό το θέμα της φτώχειας ε, και της κοινωνικής συνοχής ε, αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Ποιο θα το έλεγε αυτό ότι θα συνέβαινε στην Ευρώπη, αλλά σε κάποιε χώρε τη Νότια Ευρώπη έχει αποκτήσει διαστάσει. και μάλιστα τρομακτικέ πολλέ φορέ. Οπότε καλό είναι, είναι και επίκαιρη η έκθεση που τη συζητούμε αυτόν τον καιρό. Εμείς στην Επιτροπή μας συμφωνούμε πέρα από πολιτικές ομάδες, το είπε και ο Ανδρέας Φαμπ, ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζονται σημαντική υποστήριξη αλλά και κίνητρα από πλευράς μας για να μεταξελιχθούν. 11 εκατομμύρια είναι οι απασχολούμενοι στην Ευρώπη, 6% του συνόλου της απασχόλησης. Δεν είναι καταφρόνητη αριθμή, είναι σημαντική. Και επειδή η κρίση αυξάνεται και γίνεται τι; σε πολλές χώρες, ε, είναι σημαντικός παράγον. Συμφωνήσαμε σε κάποιες συμβαστικές τώρα τροπολογίες και χαίρομαι γι' αυτό και χαίρομαι που αναφέρεται και απαιτείται μείωση της γραφειοκρατίας γιατί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά αντιμετωπίζουν τεράστια γραφειοκρατία, ίσως και περισσότερη από άλλες επιχειρήσεις και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν οποιαδήποτε ε, διοικητικά εμπόδια να αρθούν. Και ουσιαστικά όμως και πραγματικά. Γιατί χάνουμε ε, για την εσωτερική αγορά. Και επίσης το θέμα των ε, δημοσίων συμβάσεων που μας απασχολεί. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται καλύτερη η συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων. Χρειάζεται το σωστό μείγμα απλούστευσης και συγχρονισμού. Αυτό τα λέει και η έκθεση του κυρίου Ταραμπέλα. χρειάζεται και σε αυτό κάποια βελτίωση, αλλά εργαζόμαστε παράλληλα στην Επιτροπή μας. Θέλω να τονίσω το εξής όλο, ε, όλος ιδιαίτερος, ε, την διασυνορική συνεργασία κοινωνικών επιχειρήσεων. Και εκεί υπάρχει πολύ χώρος ακόμα για συνέργειες που δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια όπου η διασυνορική συνεργασία αφορά τρεις χώρες. Είναι το τριεθνές ε, ε, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Γερμανία. Και βλέπω ακριβώς ποια είναι τα εμπόδια, ακριβώς για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Και χαίρομαι που η, η συγκήτρια ασχολείται με αυτό το θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας και το υποστηρίζει στην τροπολογία της στη συμβαστική. Εδώ ένα πάρα πολύ καυτό θέμα είναι το ζήτημα ε, της ε, υγειονομικής περίθαλψης. Με την ε, οδηγία αυτή, ως Κοινοβούλιο ανοίξαμε το δρόμο για καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και περίθαλψη. Πολλές κοινωνικές ε, επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ακριβώς σε αυτό το τομέα και θα πρέπει να βασιστούμε στην ήδη υφιστάμενη οδηγία για να ε, δημιουργήσουμε το σωστό δυναμικό. Ακριβώς σε αυτόν τον πολύ μικρό τομέα ε, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η σημασία της εσωτερικής αγοράς και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ για να ε, καταπολεμήσουμε και να ξεπεράσουμε την κρίση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους ε, συναδέλφους που με ακούσαν. Ευχαριστώ. Κύριε Ρούλε, σύντομη θα είμαι εγώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Χάντλε και έστω και εν απουσία της. Είναι καλή η βάση και η πρότασή της και πολύ επικοδομητική πάντα η συνεργασία της. θα υπερψηφίσουμε τελικά τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν συμμετείχαμε στην εκπόντιση εντατικά, γιατί είναι γνωμοδότηση και επίσης είμαστε μικρή ομάδα και πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας κάθε φορά. Θέλω επ' ευκαιρία να αναφέρω κάτι σημαντικό ε, για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν είναι όλες οι ίδιες. Υπάρχουν μικρές δομές, ε, μη ε, κερδοσκοπικές, φιλανθρωπικές, αλλά υπάρχουν και μεγάλες εμπορικές εταιρείες κοινωνικές. Και αν δεν το λάβουμε υπόψη, αυτό είναι πρόβλημα. Προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα να εξαιρούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις όταν πρόκειται ε, για τη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων ε, σε συνεργασία μεταξύ ε, ε, δύο δημοσίων φορέων. Δεν είναι σδίτ αυτό όταν συμμετέχει μια κοινωνική επιχείρηση σε συνεργασία με το δημόσιο. Δεν θεωρείται ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να είναι φιλανθρωπική ας πούμε ή μη κερδοσκοπική σε μερικές τροπολογίες έχω την άποψη ότι μπερδεύονται τα πράγματα, αλλά θα τα δούμε αυτά στις ψηφοφορίες και θα τα διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, κύριε Μακλάκη. Um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ ότι η κυρία Χάνσλικ και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις συμβιβασμού που έχουν υποβληθεί. Σε μια τροπολογία υπογράμμισα την σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είπα ότι απαιτείται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και χαίρομαι που αυτό υποστηρίζεται στην πρόσφυγη από τον εισηγητή μου με βρίσκει σύμφωνη ο εστιασμό στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι αντιμετωπίζουμε και τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ και με τι προτάσει μικροπιστώσεων για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στα πλαίσια τη πρωτοβουλία κοινωνική επιχείρηση τέθησαν ορισμένα θέματα, αλλά είμαι υπέρ της πρότασης να χρησιμοποιηθούν μικροπιστώσεις για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και χαίρομαι που και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί στο συμβιβασμό. Πολύ φοβάμαι ότι ορισμένε από τις τροπολογίες για τις δημόσιες συμβάσει δεν θα, δεν θα τύχουν τη υποστήριξη της ομάδας μου. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ε, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις. Βρήκαμε μια ε, λογική λύση, η οποία καλύπτεται από την τροπολογία 5. Σε ό,τι αφορά άλλες τροπολογίες, πιστεύω ότι οι μερικές από αυτές ε, παρέμειναν στα πλαίσια του ε, δικαίου απασχόλησης. Βεβαίω, οι χώρε μέλη είναι εκείνε που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το δίκαιο εμείς θα το στηρίξουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνούμε με το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης και τις συμβιβαστικέ προτάσεις, με εξαίρεση τη συμβιβαστική πρόταση 4. Good. Thank you. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως κάποιο άλλο μέλος θα ήθελε να πάρει μέρος στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής θα μπορούσε να κλείσει τη συζήτηση, αλλά δεν το βλέπω εδώ. Όχι. Εντάξει. Ωραία. Εξ ονόματός του και τη απουσία του, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την συμβολή του. Η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο. Η κυρία Χάνσλικ θα το προετοιμάσει. Θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο, από ό,τι κατάλαβα, η Επιτροπή Απασχόληση θα ειδωτήσει στι 10 Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αύριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο από την Επιτροπή που δεν θα να πάρει το λόγο. Όχι. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Είμαστε λίγο μπροστά από άποψη χρόνου. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε στις 11 και 4 εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Αν συμφωνείτε, θα έλεγα μέχρι τις 11 και 4 να κάνουμε το, ένα διάλειμμα και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.

Uh, so, Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 και 4, η προβλεπόμενη ώρα για να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας για δύο πολύ σημαντικές προτάσεις αφορούν την ε, καταναλωτικές διαφορές και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Κινούνται παράλληλα αυτά τα δύο, ε, αυτά τα δύο θέματα γιατί συνδέονται άμεσα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γκρέκ. Η Ρόζα Τούν δεν είναι ακόμα εδώ. Έχουμε και μερικούς σκιώδεις ηγητές, ο κύριος Άντρος, ο κύριος Ρέπο δεν είναι εδώ, ο κύριος Ρόσφορ είναι εδώ, κάνει και τις δύο εκθέσεις και ο κύριος Φόξαν και τα δύο. Χαίρομαι ιδιαίτερα να καλωσορίσω την επίλεκτη ομάδα από τη Γενική Διεύθυνση η κυρία Μαρία Κριστίνο Ρούσο, γνωστές φίλες της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων. Θα απαντήσουν λοιπόν για αυτά τα θέματα αργότερα. Δίχως άλλη καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε με τον Άλαν Μπάρκελ που θα ήθελα να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα και πώς σκοπεύουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, το σύνολο τροπολογιών ήταν 400 διαιτητικέ με 124. Οι τροπολογίε αυτέ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, αλλά οι τομεί που προκάλεσαν τι περισσότερε τροπολογίε ήταν το εύρος της πρότασης, διασυνοριακό εμπόδιο και κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία απασχολούνται από τον εμπορευόμενο. Η δεύτερη ήταν κατά πόσον οι καταναλωτέ θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με τον εμπορευόμενο πριν καταλήξουν σε μια εναλλακτική επίλυση. Το τρίτο αφορούσε την πληροφορία ότι οι πληροφορίε θα πρέπει να υποβάλουν οι εμπορευόμενοι στου καταναλωτέ. Τέταρτον, αρχέ νομιμότητα και ελευθερία. Ένα άλλα, άλλα σημαντικά θέματα κατά πόσον οι εμπορευόμενοι οι οποίοι καταγγέλνουν του καταναλωτέ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον, σε αυτό το τομέα, το κόστο τη ΕΔ και της ΕΔ ε, σε ό,τι αφορά το εύρος, νομίζω ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι οι εναλλακτικέ επιλύσει καταναλωτικών διαφορά θα μπορούσαν να, να, να αποτελέσουν μια απειλή για την αμεροληψία. Ορισμένε τροπολογίε παρόλα αυτά έχουν προταθεί. Τροπολογίε οι οποίε λένε ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό αυτό υπό τον όρο υπάρχουν ε, ε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να ληφθεί υπόψη θα δούμε μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσαμε να φτάσουμε ανάλογα με τα κριτήρια και ανάλογα με τις ρήτρε διασφάλισης που θα γίνουν δεκτές από την Επιτροπή αυτή. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει ε, να διαγράψουμε εντελώ ορισμένε ε, τροπολογίες που αφορούν ε, μέτρα διαφρύδαξη. Επίσης υπάρχουν τροπολογίες που αφορούν το δυσενεργειακό εμπόριο. Η μείωση του εύρους για την κάλυψη μόνων χώριων διαφορών θα ε, συνδημιουργήσει περαιτέρω κατακαιρματισμό και θα δημιουργήσει ένα άνισο επίπεδο προστασίας. Ορισμένες πρωτοβουλίες που προτείνουν να εξαιρεθούν ορισμένοι τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Άλλες τροπολογίες αποκλείουν πολλές υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα ε, το γενικό ενδιαφέρον μπορεί να είναι ένα ευρύτατο ε, ε, ένας ευρύτατος τομέας. Αυτό αφορά διάφορους τομείς και θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση για τους καταναλωτές και να περιορίσει τη χρησιμότητα της ε, εναλλακτική επίλυση. Συνεπώ, εγώ δεν αποκλείω συγκεκριμένου τομεί. Προσπαθώ να διευκρινίσω αυτό που θα καλύψει η οδηγία. Ε, ενοχικές ε, διαμάχες με στόχο να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο ε, εναρμόνισης. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες των χωρών μερών για να δούμε αν υπάρχει αντίφαση με το εθνικό δίκαιο. Το δεύτερο, ο κύκλος ε, τροπολογιών αφορούν την υποχρέωση των καταναλωτών να ενημερώνουν τον εμπορευόμενο. Συμφωνώ ότι σε γενικέ γραμμέ ε, πριν καταφύγουν στην επίλυση διαφορών, οι καταναλωτέ θα πρέπει να ενημερώνουν τον εμπορευόμενο. Σε βάση ορισμένων τροπολογιών αυτό είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε του καταναλωτέ να επικοινωνούν με τον εμπορευόμενο, αλλά να του αφήσουμε τη διακριτική ευχαίρεια κατά πόσο θα καταφύγουν στο δικαστήριο, όπω αναφέρεται από τη χάρη θα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στην τροπολογία μου αναφέρομαι στην αρχή ότι χώρες μέλη θα μπορούσαν να διατηρήσουν τους διαδικαστικούς κανόνες εναλλακτική επίλυσης που επιτρέπουν στους φορείς εναλλακτική επίλυσης να λειτουργήσουν περισσότερο αποτελεσματικά μόλις υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας. υποχρέωση του καταναλωτή να επικοινωνήσει με τον εμπορευόμενο πριν καταφύγει στην εναλλακτική επίλυση είναι ένα διαδικαστικό κανόνα που υπάρχει σε ορισμένε χώρε μέλη, αλλά όχι σε όλε. Διευκρινίζοντα ένα τέτοιο διαδικαστικό κανόνα, ε, θα ε, τον προωθήσουμε και στις 27 χώρες μέλη, πράγμα που δεν είναι αναγκαίο. Όπως είπα σε αυτή την οδηγία, στόχο έχουμε να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση της ε, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για την ποιότητα της εναλλακτική επίλυσης. Οι διαδικαστικοί κανόνες είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Υποχρέωση ενημέρωση. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες ε, τροπολογίες μας δείχνουν ότι ο εμπορευόμενο θα πρέπει να δώσει στου καταναλωτές ορισμένες πληροφορίες. Μερικές από τις τροπολογίες που λάβαμε περιορίζουν σοβαρά τις ε, παροχή πληροφοριών και πάλι συνεπώ, πιστεύω ότι αυτό που θα αποδυναμώσει του καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία και την νομιμότητα, μία σειρά από βουλευτές ε, υπέβαλαν τροπολογίες ε, για την ελευθερία και την νομιμότητα. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε γραμμέ, γραμμές, τροπολογίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και συνεπώς δεν θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ένα συμβιβασμό και στις δύο αυτές αρχές. Το πέμπτο θέμα που αποφάσισα ότι θα είναι σημαντικό είναι ε, αφορά τους εμπορευόμενους που στρέφονται κατά το καταναλωτών. Ορισμένες ε, ε, τροπολογίες επιτρέπουν στους εμπορευόμενους να το κάνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η εναρμόνιση σε αυτό το σημείο θα είναι αντιπαραγωγική. Θα πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση των επιπτώσεων και από το feedback που άκουσα δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που να θέλουν, που να χρειάζονται ένα τέτοιο εργαλείο. Συνήθω το μοναδικό παράπονο που έχουν οι εμπορευόμενοι είναι η μη πληρωμή. Υπάρχουν άλλες, ε, άλλα προβλήματα, είναι περιορισμένα και κατά συνέπεια δεν ε, ε, είναι τα πλέον κατάλληλα για εναλλακτική επίλυση. κόστο συμμετοχή. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις τροπολογίες που αναφέρονται ότι ε, ο, αυτός που έχει χάσει την υπόθεση θα πρέπει να αποζημιώσει. Αυτό θα είναι αποτρεπτικό για τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική επίλυση. Επίση όμω εναρμονίζει και τον τρόπο λειτουργία των φορέων. Δεν είναι στόχο αυτό τη οδηγία. Συνεπώ, συμφωνώ με την άποψη ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν για του καταναλωτέ και ότι η μορφή χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών ανεξαρτησία. Συμπεριέλαβα την αρχή της ανεξαρτησίας το σχέδιο έκθεσης ως ξεχωριστό άρθρο, αλλά λάβαμε αρκετές τροπολογίες για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία. Προσπάθησα να γράψω ένα συμβιβασμό με, με τις δύο ε, αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις. Συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, οι δικοί μας μας απόψεις ταυτίζονται σε μία σειρά από θέματα, αλλά κυρίω την ελευθερία και την νομιμότητα. Αλλά υπάρχουν ορισμένες αναντιστοιχίες ό,τι αφορά την παρογή πληροφοριών και το, εύρος, και το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Ένα θέμα που θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια των τριμερών συζητήσεων. Έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση για τις 28 Ιουνίου. Θα ήθελα όμως τώρα να ακούσω τα σχόλια από τους συναδέλφους και από τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα πρότεινα, επειδή υπάρχουν μερικοί κοινοί σκιώδει εισηγητέ, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Τούν, η οποία είναι εισηγήτρια για την ε, ε, οδηγία και μετά μπορούν να πάρουν το λόγο και οι σκιώδεις εισηγητές. Να γίνει το ένα μετά το άλλο. Μόνο κύριος, κυρία Γκέτμαρ, εσείς θα πάρετε το λόγο για τον κύριο Ρέπο. Μάλιστα. Κυρία Τούν, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω στα αγγλικά. Συναντήθηκα αρκετές φορές με τους Σκιώδης και σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις τροπολογίες. Αυτό μας βοήθησε ιδιαίτερα και είχα και συναντήσει με την Επιτροπή, με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής σε σχέση με την εναλλακτική επίλυση διαφορών, ηλεκτρονική επίλυση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, ίσως όχι τώρα, work Και θα μας απασχολεί στην Ευρώπη όπως και όπως ισχύει και για το Solvit και άλλα σχέδια. Έλαβα πολλές τροπολογίες. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι όταν ακούσαμε την εισήγηση του κυρίου Γκρέχ βλέπουμε ότι η ηλεκτρονική επίλυση θα πρέπει να αφορά ένα ξεχωριστό θέμα, ένα επιμέρους θέμα. Ο καταναλωτής ή ο έμπορος υποβάλλει αυτή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών έτσι ώστε να επιληθούν διαφορές στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ηλεκτρονική επίλυση αφορά την ε, εξαγγελία της, αφορά την καταγγελία η οποία στη συνέχεια εντάσσεται στο ADR, στην εναλλακτική επίλυση διαφορών. Έλαβα αρκετές τροπολογίες. Μία που είναι αρκετά σημαντική και με βρίσκει σύμφωνη αφορά το εξής. Αν πρόκειται για επιγραμμική υπόθεση, η φυσική παρουσία του προσώπου δεν είναι απαραίτητη. Συμφωνώ απόλυτα. Υποβλήθηκε από αρκετού συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για ε, πρόσωπα, για διευκόλυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επίλυσης. Μίλησε για facilitators μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επίλυσης και πολλοί από εσάς ε, εκφράστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Μιλήσατε για απαλυφή. Πρόκειται για επικάλυψη, διότι ήδη έχουμε ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και σημεία ε, συνάντηση, σημεία ηλεκτρονικής ε, επίλυσης διαφορών. Άρα δεν θα πρέπει να γίνει λόγος ειδική μνήμα για τους facilitators. Έλαβα πολλές αρκετές τροπολογίες που σχετίζονται με την εναλλακτική επίλυση διαφορών με το ADR γενικότερα. Πρότεινα να μην υπάρχει σύγχυση, δηλαδή το ODR, η ηλεκτρονική επίλυση, αφορά ένα ειδικό πλαίσιο επίλυσης διαφορών και δεν πρέπει να ενταχθεί στο ADR, γενικότερα στην εναλλακτική επίλυση διαφορών, τη μη ηλεκτρονική. Το κείμενο πρέπει να διασαφινιστεί κάπως. Προσπάθησα να αποβάλω ό,τι δεν είναι αναγκαίο, ό,τι πλεονάζει. γιατί ήθελα να απλουστευτεί η όλη διαδικασία. Γι' αυτό πρότεινα το μέρος που θα επιλέξει το ADR, δηλαδή την εναλλακτική επίλυση, ε, να, πρέπει να ανταποκριθεί, να είναι και ο ανταποκρινόμενος. Θα ήθελα μία διασάφηση από την Επίτροπη, γιατί μιλάμε για καταναλωτή προς επιχείρηση, αλλά και επιχείρηση προς καταναλωτή. Αυτό αυτό είναι ύψης της σημασίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Έγιναν διαβουλεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ε, διοργάνωσα κάτι τέτοιο και το 75% των απαντώντων είπε ότι χρειάζεται μέσα στα πλαίσια της επιγραμμικής αντιστάθμισης ή αντικαταβολής. Άρα ε, οι απαντώντες ή ανταποκρινόμενοι είναι επιχειρήσεις ή καταναλωτές, αλλά κυρίως είναι έμποροι, γι' αυτό θα πρέπει να ενταχθούν στο ADR, στην εναλλακτική επίλυση διαφόρων. Οι σκιώδεις εξέφρασαν μία επιθυμία και συμφώνησα κι εγώ Ζητήσαμε ε, μεγαλύτερη προθεσμία για την επιλογή του ADR για τον ας πούμε ε, ενάγοντα και εναγόμενο 20 ημέρες δηλαδή και για το ODR και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα βασικά ζητήματα διαφορών Πολύ ζητήσατε το ODR, η ηλεκτρονική επίλυση, να αφορά καταναλωτές κατά επιχειρήσεων, αποκλειστικά. Αυτό θα το συζητήσουμε. Μετά έγιναν συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς θέματα μετάφρασης. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα μεταφράσεων, δηλαδή ε, μηχανογράφηση και ανθρώπινος ε, παράγων, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Πολλές διαβουλεύσεις έγιναν και πιστεύω ότι η επίλυση, η, ε, η μετάφραση και η ευθύνη για τη μετάφραση θα πρέπει να ισχύει σε ένα σημείο. Ένα άλλο θέμα ήταν η προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχουμε μία ιστοσελίδα, μία ηλεκτρονική πύλη και εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκή ηλεκτρονική τότε η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να απαιτήσουμε από τους καταναλωτές να μάθουν άλλες μορφές πρόσβασης. Αν θέλουμε να απλουστεύσουμε τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μία διεύθυνση όπου ο καταναλωτής θα βρίσκει τα πάντα. Να έχουμε μία δηλαδή ηλεκτρονική πύλη και όλα να εντάσσονται σε αυτή την πύλη και να υπάρχει άμεση πρόσβαση και από άλλες ιστοσελίδες. Αυτό από τεχνικής πλευράς είναι πολύ εύκολο. Όλα λοιπόν να εντάσσονται σε μία δικτυακή πύλη. Την επόμενη εβδομάδα με τους Σκιώδης θα συζητήσουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού στις 9 Ιουλίου είναι προθεσμία και θα ψηφίσουμε στις 10 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις, τη δική σας συνεισφορά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και για τη δική σας ε, ηγεσία στη προσπάθεια αυτή και για την κατεύθυνση που δίνετε. Γιατί έχουμε αρκετές τροπολογίες και για τις δύο εκθέσεις έχετε συζητήσει για τροπολογίες που θεωρείτε πιο κατάλληλες ε, για την έκθεση του Λουί Γκρέχ. Δηλαδή εκεί πρέπει να κατατεθούν και όχι στη δική σας έκθεση. Θα πρέπει να το δείτε αυτό διμερώς. Ας έρθουμε τώρα λοιπόν στους Σκιώδης. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα με την εξή σειρά. Μάιερ. Σκιώδης ε, για την ADR, την εναλλακτική επίλυση από το ΕΛΚ η κυρία Γκέπχαρτ που θα μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Ρέπο για την ηλεκτρονική επίλυση, ο κύριος Ροσφόρ, Ρούλε και Φόξ και για τις δύο και ο Ντένις Δε Γιόγκ που τον καλωσορίζω. Βλέπω και εσύ Ντένις καλύπτεις και τις δύο εκθέσεις. Ωραία. Ο Χάντς Πέτσα Μάια. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πάνω από 400 είναι οι τροπολογίες και τι δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα και πόσο σοβαρά το παίρνουν υπόψη οι συνάδελφοι. Και εγώ στο μεταξύ είχα συνομιλίες με τον εισηγητή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστώθηκε ότι κάθε φορά που οι ε, τροπολογίες δεν είναι σίγουρο που ανήκουν θα πρέπει να ξέρουμε ότι ήδη σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ διαφορετικά συστήματα που ισχύουν όμως ήδη. Και αυτά θα πρέπει να συνδεθούν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχει νόημα να εφευρίσκουμε κάθε μέρα τον τροχό και να τα ξεκινάμε από μηδενική βάση επειδή έρχεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Λοιπόν, εφόσον θέλουμε να συνδέσουμε τα υφιστάμενα συστήματα θα πρέπει κάπως να δεχτούμε και να σεβαστούμε και τις δικές τους ιδιαιτερότητες σε κάθε χώρα. Παράδειγμα, Υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις στο κείμενο που προτείνεται που μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις. Παράδειγμα, η υπηρεσία εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί να κάνει είτε πρόταση, είτε να λάβει και δεσμευτική μάλιστα απόφαση. Αυτό δεν θα πρέπει να παρεξηγηθεί ότι επειδή εμείς κάνουμε ε, νομοθεσία, ορίζουμε αν θα κάνει πρόταση ή αν θα λαμβάνει απόφαση, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν αν αυτές οι υπηρεσίες μπορούν μόνο να προτείνουν ή μπορούν και να αποφασίζουν. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα δούμε σε συζήτηση και λογικά να τα ρυθμίζουμε. Δυσκολίες τώρα έχουμε από τη γερμανική σκοπιά ιδιαίτερως αλλά και από άλλους είναι το, τα θέματα της κοινοφελής υπηρεσίας των ΔΕΚΟ γενικά ή του Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Υπάρχει η Γενική Αρχή ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών να αποφασίζουν τι χαρακτηρίζουν κοινοφελείς υπηρεσίες και τι ε, αποχαρακτηρίζουν. Εάν λοιπόν αυτό ε, ισχύει, τότε η τελική επανόρθωση και αποζημίωση δεν είναι συμβατική υποχρέωση, αλλά είναι ε, εκ νόμου. Δηλαδή, όταν έχεις ε, αξίωση που υποστηρίζεται από νόμο, δεν είναι συμβατική υποχρέωση. Υπάρχουν όμως και μικτές συμβάσεις, αλλά υπάρχει το δημόσιο συμφέρον και η υποχρέωση διανόμου ε, να ε, επανορθώνεται αυτό. Ακόμα και αν διαπληκτίζονται και τσακώνονται ορισμένοι, εφόσον υπάρχει νόμος θα πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση. Δεν έχει να κάνει με συμβάσεις και συμφωνίες κτλ. Και, και αυτό δεν ενδείκνυται για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θα πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση. Θα πρέπει, λέει, πάντα ε, να προσπαθεί κάποιος να το ρυθμίζει διμερώς για να αποφορτίζεται αυτή η υπηρεσία. Ε, καλό είναι αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που το έχουν ρυθμίσει αυτό. Δεν θα πρέπει να τα αναγκάσουμε να το αλλάξουν. Ότι οπωσδήποτε ελάτε σε επαφή με τον έμπορο. Όχι. Αφού το έχουν ρυθμίσει αλλιώ οι χώρε, πρέπει να κάνουμε εμεί μακρέ συζητήσει αν είναι θέμα επικουρικότητα ή όχι. Αν συμφωνούμε ότι τα υφιστάμενα συστήματα σε μεγάλο βαθμό πρέπει να ενσωματωθούν, θα πρέπει να πούμε και εδώ ότι τα αφήνουμε ε, στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Αλλά συνιστούμε, ακριβώς για να μην ε, επιβαρύνονται ιδιαίτερα αυτές οι θέσεις, τα σημεία ADR, να έρχονται σε επαφή εκ των προτέρων, μάλλον προηγουμένως, συγγνώμη, με τον έμπορο, μήπως λεχθεί το ζήτημα διαφορετικά. Τα ήδη φυστάμενα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ανεξαρτησία, ποιότητα, είναι απόλυτες αναγκαιότητες. Ε, είναι γεγονός αυτό και σαφές, αλλά τι θα κάνουμε τώρα με κάποια συστήματα που έχουν ορισμένες εταιρείε στο εσωτερικό τους και αυτές θα τις υιοθετήσουμε τις μορφές. Είναι ανεξάρτητες, αλλά πληρούν τις απαραίτητες ποιοτικέ απαιτήσεις. Στη Γερμανία, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, ακόμα και ένας δικηγόρος που ε, παρίσταται στο δικαστήριο και θα πρέπει να είναι απολύτως ε, ανεξάρτητος, μπορεί να είναι υπάλληλο μιας εταιρείας αλλά θα πρέπει η εταιρεία γραπτός να ορίσει ότι έχει τη ελευθερία ο δικηγόρος όταν υπάρχει πρόβλημα να το κάνει με ανεξαρτησία και με δική του ευθύνη και συνείδηση. Και αυτά τα θέματα θα πρέπει ενδεχομένως να τα δεχτούμε. Για το κόστος τώρα. Δωρεάν, φθηνά, δεν ξέρω τι άλλο προτείνει ο εισηγητής. όταν χάσει την υπόθεση ο καταναλωτή θα πρέπει να πληρώνει. Όχι, να το πούμε διαφορετικά. Ένα μικρό κατόφλι να υπάρχει δεν πειράζει ε, για να μην προκαλέσουμε και γενικό πανικό να τρέχουν όλοι να ζητάνε. Λοιπόν, ε, και ε, όταν κάτι είναι δωρεάν δεν βλάπτει κιόλα, αλλά να μην πληρώσει ο καταναλωτής. Το αντίθετο, όταν κερδίζει να παίρνει τα χρήματά του πίσω. Είναι διαφορετική η προσέγγιση από την αρχή. Να πει ο καταναλωτής, ότι μπαίνω ε, στο ρίσκο, παίρνω το ρίσκο να, να πληρώσω 30 ή 50 ευρώ, αλλά αν κερδίσω τα πάρω πίσω. Και όχι ε, ότι μπαίνω ε, στον κίνδυνο να πληρώσω ένα οποιοδήποτε κόστος προκύψει που δεν μπορώ καν να το επηρεάσω για απόφαση εις βάρος μου. να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό που να καταβάλει ω εγγύηση, α πούμε, ο καταναλωτή και όταν δικαιωθεί να το παίρνει πίσω. Αυτό είναι νομίζω καλύτερη λύση. Το θέμα τώρα, αν μπορεί μόνο ένας καταναλωτής να προσφύγει για εναλλακτική επίλυση διαφορών ή και ένας επιχειρηματίας. Ποιο είναι ο στόχος, να είναι εξοδικαστική η ρύθμιση, να μην πάμε στα δικαστήρια. Δηλαδή θεωρητικά θα μπορούσε και η επιχείρηση να τηλεφωνήσει στην εναλλακτική επίρρηση διαφορών. Τώρα κατά πόσο γίνεται αυτό στην πράξη είναι άλλη ιστορία. Συνήθως οι επιχειρήσεις δεν ζητούν αποζημίωση, ή επανόρθωση, αλλά ανάκτηση των χρημάτων. Δηλαδή μπορεί να έχει νόημα να προσφύγουν εκεί για να πούν στον καταναλωτή φέρει τα λεφτά πίσω, αλλιώ θα σε πάω στα δικαστήρια. Αν α πούμε όμω μια καφετιέρα κάνει 90 ευρώ και ο καταναλωτή αρνείται να δώσει και τα χρήματα και την καφετιέρα, ξέρω εγώ, δεν έχει νόημα να πάει στο δικαστήριο. Εκεί μπορεί ο κατασκευαστή να απευθυνθεί στην εναλλακτική επίλυση διαφορών για να αποφευθεί και πολύ κόστο για τον καταναλωτή. Γενικά, κοιτάξαμε τι γίνεται με τη γραφειοκρατία, αν μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Καθόλου γραφειοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά υπάρχουν κάποιες προτάσεις που είναι πολύ προβληματικές. Θέλουμε όσο γίνεται να είναι απλά τα πράγματα. Γενικά πιστεύω ότι στις συζητήσεις ε, μπορέσαμε να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Ορισμένα πράγματα χρειάζονται προφορικές συμπληρώσεις ή στις συμβιβαστικές μπορούμε και να τα αλλάξουμε. Και αυτά είναι μεταφραστικά λάθη που είπε ε, η συνάδελφος. Γιατί πολλές φορές όταν είναι λάθος η μετάφραση ή η διαφορετική διατύπωση βγαίνει το αντίστοιχο νόημα. Οι μεταφράσει είναι γενικότερα πρόβλημα. Σιγά σιγά αυξάνονται τα προβλήματα, περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Λοιπόν, γενικά πιστεύω από τις 400 τροπολογίες μπορούμε τις περισσότερες να τις καλύψουμε με συμβιβαστικέ και γι' αυτό προτείνω να αφήσουμε λίγο χρόνο πώς έχει η πραγματικότητα. Την άλλη εβδομάδα φεύγουμε όλοι. Το έλκυνε στη Φινλανδία, οι σοσιαλιστές, δεν ξέρω πού πάτε εσείς, Άλλος κανείς Στρασβούργο την παραπάνω επόμενη εβδομάδα χωρίς βοηθούς, χωρίς κομισιόν. Κανονικά στις 10 του μηνό Ιουλίου δεν μπορούμε να ψηφίσουμε λογικά εκτός να ψηφίσουμε και τις 400 τροπολογίες. Το καλύτερο και λογικό είναι να ψηφίσουμε μέσα Σεπτεμβρίου με λιγότερες συμβιβαστικές πλέον τροπολογίες οπότε ας τα κάνουμε σωστά και με την ησυχία μας αυτά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της προθεσμίας θα πρέπει να συζητηθεί από εισηγητή και σκιώδης και θα το δουν και οι συντονιστές αύριο το απόγευμα το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Μπορείτε να το θίξετε τώρα. Η κυρία Γκέπχαρτ τώρα θα μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου ε, Ρέπο σε σχέση με την ηλεκτρονική διευθέτηση διαφορών. Ευχαριστώ. Με παρακάλεσε ο κύριος Ρέπο να τον εκπροσωπήσω σήμερα διότι δυστυχώς έπρεπε να πάει σε μια κηδεία ενός πολύ καλού του φίλου και ε, δεν μπορούσε να είναι στις Βρυξέλλες, μου άφησε όμως ένα σημείωμα. Για την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, ο κύριος ε, Ρέπο ε, ε, συμφωνεί, επενεί την εισηγήτρια, η οποία και το αξίζει. του αρέσει ιδιαίτερα η τροπολογία υπαριθμών 6 του κυρίου Ρέπο, όπου προτείνεται ε, να επιτρέπεται σε όλους τους καταναλωτές και τους εμπόρους να υποβάλουν τις καταγγελίες τους συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροπολογία 6 τα λέει αυτά. Αυτό ε, απλουστεύει τρομερά όλη τη διαδικασία. Επίσης, του αρέσει πολύ η ιδέα της τροπολογίας υπαριθμών 21 ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι δωρεάν, χωρίς χρέωση λέει εδώ. Επίσης θεωρεί πολύ σωστό αυτό που λέει η τροπολογία υπαριθμών 57 για την προθεσμία ε, των 30 ημερών που ζητάει η τροπολογία να διαγραφεί αυτό. Και γενικά συμφωνεί με την έκθεση. Έχει όμως ένα πρόβλημα με την τροπολογία υπαριθμών 29 όπου αναφέρονται οι μεταφράσεις. Δηλαδή ποιος είναι αρμόδιος και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και πώς λειτουργεί. Οπωσδήποτε να το κοιτάξει αυτό. Και δεν, ε, του αρέσει και η τροπολογία σας υπαριθμών 86. Διότι Όταν υπάρχουν αυτόματες μεταφράσεις που τις κάνουν με μηχανήματα, είναι προβληματικό. Γιατί οι πολίτες δεν κάνουν τις καταγγελίες τους σε μία γλώσσα πολύ καλά διατυπωμένη. Πολλές φορές χρησιμοποιούν διάλεκτο, σλάνγκ και το μηχάνημα δεν το καταλαβαίνει, μεταφράζει άλλα αντάλλων και υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Πώς ε, θα αντιμετωπιστεί. Ο κύριος Ρέπο έχει κάνει και αυτό τροπολογία στο θέμα της προθεσμίας. Δηλαδή, μέσα σε ποιο διάστημα θα πρέπει να δίνεται η απάντηση σε μια καταγγελία, ένα παράπονο. Και θεωρεί ότι αυτό που προτείνεται εδώ, 30 ημέρες αν δεν απατώμε, είναι προβληματικό. Διότι μέσα σε ένα μήνα συμπεριλαμβάνεται και η συγκέντρωση των εγγράφων. Ε, δηλαδή μειώνεται έτσι η, ε, το διάστημα που ε, υπάρχει για τη λήψη της απόφασης. Πάντως γενικά πιστεύει ότι μπορεί να είναι καλή συνεργασία με την εισηγήτρια γιατί συμφωνεί με τις περισσότερες τοπολογίες της Ρόζα. Η τοπολογία του κυρίου Ρέπο είναι 254. Ε, ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, let's move on. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ροσφόρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ τους δύο εισηγητές και να τους ευχαριστήσω για την εξαιρετική τους εργασία που θα έχει μεγάλη ανταπόκριση. Θα προσπαθήσω να δούμε ορισμένα θέματα. Δεν είναι δύσκολο να είμαστε σε δύο πεδία, σε δύο κείμενα, αλλά θα ήθελα να το προσπαθήσω θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός του πεδίου εφαρμογής ADR και ODR, ηλεκτρονικής και μη επίλυσης, δηλαδή σε σχέση με τις επιχειρήσεις και του καταναλωτή. Είμαι της άποψης του κυρίου Γκρές ότι θα πρέπει κατά κύριο λόγο να μας απασχολούν οι καταναλωτές. Και όπως είπε η κυρία Τούν, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τον καταναλωτή πρωτίστως θα πρέπει να είναι ένα μέσο το οποίο να υπηρετεί τους καταναλωτές. Και οι επιχειρήσεις, όπως είπε και ο κύριος Γκρέχ, δεν είναι βασικοί καταγγέλλοντες. Μερικές είναι, αλλά όχι πολλές. Άρα και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με εναλλακτικά μέσα επίλυσης διαφορών ε, online και να μιλάμε για πλαίσιο consumer to business. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Το πιο σημαντικό θέμα, όπως υπενθύμησαν πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μάιερ, αφορά τον διαμεσολαβητή επιχειρήσεων. Οι δικές μου επιχειρήσεις άπτονται αυτού του θέματος, γιατί θα πρέπει να ενσωματώσουμε στο σύστημα αυτό, αυτά που προϋπάρχουν δηλαδή τους διαμεσολαβητές επιχειρήσεων που υπάρχουν σε αρκετές χώρες. Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν από συναδέλφους και ιδιαίτερα τους Γάλλους, ένας εκ των οποίων με κοιτάει στα μάτια αυτή τη στιγμή, αφορούν την ασφάλεια, το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, την ανεξαρτησία και ε, είναι σαν να προβάλλουμε ένα συνικό τείχος δηλαδή, μεταξύ του διαμεσολαβητή και, εκείνης, και της επιχείρησης της ίδιας και ενός αναγνωρισμένου καταναλωτή. Εδώ γίνεται μία ετήσια αποτίμηση από μία ανεξάρτητη αρχή, κάτι το οποίο είναι άκρος αποτελεσματικό. Περνώ από το ένα κείμενο στο άλλο γιατί πρέπει να εργαστούμε επί των δύο. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής επίλυσης δεν υπάρχει άμεση διαμεσολάβηση με ένα φυσικό δηλαδή πρόσωπο, αλλά γίνεται ηλεκτρονικά. Κατανοώ τα σχόλια της κυρίας Τούν για τους διαμεσολαβητές και γνωρίζω ότι δεν είναι πάντα εύκολο να κινητοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι διαμεσολαβητές. Αλλά δεν μπορούμε να τους ε, διαγράψουμε, να τους απαλείψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τη λέξη facilitators. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαμεσολαβητές, αλλά να έχουν ε, βοηθητικό καθαρά ρόλο όταν ε, τους χρειάζονται οι καταναλωτές. Ως προς το θέμα της ηλεκτρονικής επίλυσης, θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που δεν αναφέρθηκε. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων. Γιατί όταν μπαίνουν σε ιστοσελίδες προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να την χάνουν προστασίες. Τάσομαι υπέρ της ιδέας της ειδικής, μιας ειδικής πλατφόρμας για τις ε, ηλεκτρονικές επιλύσεις, κάτι σαν το Yuri Europe. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζητάμε από την Επιτροπή συγκεκριμένες εγγυήσει και διευκολύνσεις ως προς τις πλατφόρμες. Ζητάμε επικαιροποίηση, μεταφράσεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία ειδική ιστοσελίδα για τις ε, ηλεκτρονικές επιλύσεις διαφορών με διασφάλιση προσωπικών δεδομένων. Μιλήσαμε για περιορισμό του πεδίου εφαρμογής και θα ήθελα να πω ότι οι τροπολογίες του κυρίου Φόξ με βρίσκουν σύμφωνο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τις εντάξουμε η εισηγήτρια θα ασχοληθεί με τις τροπολογίες συμβιβασμού που είναι απαραίτητες. Ως προς το κείμενο Γκρέχ, γιατί κινούμε ανάμεσα στα δύο κείμενα, θα ήθελα να πω ότι πριν ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει το ADR, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους ε, εμπόρους, με τον επαγγελματικό κλάδο. Ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πάντα. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να γίνει μια επαφή με την επιχείρηση, να υπάρχουν επαφές πριν την προσφυγή στην ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών, να υπάρχει ένα σχήμα ευελιξίας. Να υπάρχει μια προτροπή του καταναλωτή ώστε να επιληθεί το ζήτημα πριν καν προσφύγουμε στο ADR. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα διαφάνειας που δεν είναι εύκολο ως ε, προς την ηλεκτρονική υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν εύκολα κάπου. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Ως προς το κόστος τώρα, θα ήθελα να το προσεγγίσω κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση του καταναλωτή και τα κράτη-μέλη να οργανώνουν τα... το σχήμα αυτό κάπως διαφορετικά. Αλλά μία εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν σημαίνει ότι ένα συμβαλόμενο μέρος ε, ε σφάλει και το άλλο όχι. Δηλαδή δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καταναλωτής σφάλει ή η επιχείρηση σφάλει 100%. Και τη στιγμή που η δαπάνη αναλαμβάνεται από το συμβαλόμενο μέρος που σφάλει, ε, δεν έχουμε δίκιο να το αναφέρουμε έτσι, γιατί ε, τα ADR βασίζονται σε, καθαρά, σε σχήματα πολιτικής ε, δικονομίας και δεν είναι σωστό αυτό. θα πρέπει να προβάλλουμε ένα εναλλακτικό σχήμα, πιο ευέλικτο, πιο συμφιλιωτικό και να μην προβάλλει μία διαδικασία όπως ισχύει στα δικαστήρια, μία διαδικασία κατά αντιμολία. Θα πρέπει να αποκλειστεί η υγεία και τα εθνικά συστήματα υγείας και θα πρέπει να μιλάμε και για τις μη οικονομικές υπηρεσίες στα πλαίσια των ΔΕΚΟ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον καλό δρόμο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και ως προς τις τροπολογίες. Λοιπόν, σας... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν ήθελα όμως ε, να πιέσω την Επιτροπή και να πάρει το λόγο στο τέλος. Ξέρω και η κυρία Ρούλα σέβεται πάρα πολύ το χρόνο που έχει στη διάθεσή της. Παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να πω ότι έχει ε, δίκιο ο κύριος Μάγερ για τις συμβαστικές τροπολογίες να τις δούμε με την ησυχία μας και να συνεννοηθούμε. Γιατί πιστεύω ότι πολλές ε, τροπολογίες ε, φέρουν τη σφραγίδα της εθνικής εμπειρίας που έχει ο καθένας στη χώρα του. Λοιπόν, να κοιτάξουμε ξανά όλες αυτές τις τροπολογίες, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση που να οδηγήσει σε μια εναρμόνιση και να σέβεται όμως τις εθνικές ιδιαιτερότητες χωρίς να τις προσβάλλει. Αυτό είναι το ένα. Ένα άλλο σημείο που θέλετε ιδιαίτερη προσοχή είναι το πεδίο εφαρμογή. Τι θα πρέπει να εντάσσεται εκεί. Και αυτά που είπε ο κύριο Μάγερ και αυτά που είπε ο κύριο Ροσφόρ τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Να πούμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω εκεί ε, δεν ε, τα έχει διευκρινίσει αρκετά. Και το θέμα του κόστου, και η τελευταία μου παρατήρηση, έχει δίκιο ο κύριο Ροσφόρ το θεωρώ προβληματικό. Εάν καταρχήν αυτό το σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ε, κυριαρχείται από την ιδέα του κόστους. Γιατί ε, και αν είναι κόστος της τάξεως της δίκης. Εάν ο καταναλωτής θεωρήσει ότι δεν έχει πλέον εκτήματα γιατί είναι πολύ ακριβό, δεν θα το χρησιμοποιήσει καθόλου. Ε, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή να του βγαίνει πιο ακριβό από το δικαστήριο, αλλά εάν κερδίσει ε, να πρέπει να το αποζημιώνουν το κόστος, δεν ξέρω. Έχω μια ερώτηση στον κύριο Ροσφόρ, μήπως είναι θέμα μετάφρασης. Θέλετε πραγματικά τα συστήματα διαμεσολαβητών να τα εντάξετε μέσα στη διαδικασία εναλλακτική επίλυση διαφορών. Εκεί έχω επιφυλάξει εγώ γιατί είναι διαφορετικέ οι διαδικασίε. Πώ θα βρεθεί ένα μεικτό σύστημα. Για μένα είναι πρόβλημα αυτό. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε την ε, ευκαιρία να το συζητήσετε αργότερα. Ο κύριος ε, Φόξ. Περίμενε υπομονετικά και νομίζω ότι έχει ορισμένα σημαντικά σημεία να μας αναφέρει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας είμαι ευγνώμων που δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κρέτη τα σχόλια και χαίρομαι που βρίσκεται ανάμεσά μας και υγιής. Τώρα να περάσουμε στις ίδιες τις τροπολογίες. Ο δικός μου σκοπός ήταν να προσθέσω στην πολύ σωστή δουλειά που έκανε ο κύριος Γκρέξ, έτσι ώστε οι διαφορές αυτές να μπορούν να επιλύονται με τρόπο άτυπο και ταχαίως. Ένας άλλος στόχος των τροπολογιών είναι το να υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι αποτελεσματικά και θα γίνονται σεβαστά. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε, να κυρώσουμε όσα λειτουργούν πολύ καλά και πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ το να ε, <clears throat> περιορίσουμε αυτό από το B. Οι μηχανισμοί EDR, ηλεκτρονικής επίλυσης, υπάρχουν για να επιδιορθωθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των εμπορευόμενων και καταναλωτών. Εγώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα παράπονα των καταναλωτών. Χαίρομαι που μπορώ να συμφορήσω με τον κύριο Γκρέ και τον κύριο Ρόσφο ότι οι διαδικασίε του ADR θα πρέπει να είναι δωρεάν για του καταναλωτέ. Οι καταναλωτέ θα ε, δεν θα χρησιμοποιούν το μηχανισμό αυτό εάν αυτό συνεπάγεται κάθε δαπάνη. Και δεν πιστεύω πιστεύω ότι το να είναι δωρεάν το σύστημα θα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να το χρησιμοποιεί κανείς για πίδημα. Για... Θα πρέπει λοιπόν να διαβρίσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης από την βιομηχανία και θα έλεγα να γίνει μια προσπάθεια συμβιβασμού σε, αυτή την περι... σε αυτό το τομέα. Χαίρομαι που υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ, έτσι ώστε στο πεδίο εφαρμογής να, συμπεριλαμβα... να συμπεριληφθούν εσωτερικές διαδικασίες διαβεσολάβησης υπό την όρο. Υπάρχουν ρήτρες που διασφαλίζουν την αμεροληψία. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με τον κύριο Κρακέ. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου τώρα να, να ασχοληθώ στο... στην έκθεση της κυρίας ε, την ηλεκτρονική ε, επίλυση. Οι τροπολογίες μου θέλουν να διασφαλίσουν το ότι δεν θα παραπλανηθούν ή δεν θα, έχουν, ε, δεν θα τρέφουν ε, φρούδες προσδοκίες οι καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τους διαμεσολαβητές, Πιστεύω ότι αυτό συνεπάγεται μία επικάλυψη. Θα ήταν σκοπιμότερο τα σημεία, να υπάρξουν τα σημεία επαφής και οι χώρες μέλη να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Επίσης θα ήταν θετικό για τους καταναλωτές να διευκρινίσουν τι είδου βοήθεια θα πρέπει να παράσχεται. Θέλουμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής ε, ε, επίλυσης ενημερώνει για την εναλλακτική επίλυση. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένω τη συνεργασία με την κυρία Τούν και τους σκιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Για να τελειώσουμε τώρα με τον κύκλο των σκιωδών εισηγητών, ο κύριο Ντιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος της ομάδας μου στην κυρία Τούνε, διότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και μου άφησε και εμένα ένα έγγραφο να το διαβάσω. Αλλά ε, πολύ σύντομα θα καλύψει ε, την χρονική διαφορά και την εστέρηση και θα έρθει και θα συνεργαστεί. Θα περιοριστώ στην έκθεση του κυρίου Γκρέγ για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαν ε, Ντεκάμπ ε, του ΕΛΚ, ε, το συμπατριώτη μου, για την πολύ καλή συνεργασία. Μας προσέγγισαν και ανέμποροι στην Ολλανδία, αλλά και οργανώσεις καταναλωτών και τους δύο. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα στην Ολλανδία για το λιανεμπόριο που δεν πρέπει να αποκτήσει προβλήματα λόγω ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Είναι ένα σύστημα εθελοντικό και είναι πανευτυχής και οι έμποροι και οι καταναλωτές. Γι' αυτό έχουμε κάνει τροπολογίες που φιλοδοξούν στο να διατηρήσουμε το υφιστάμενο στην Ολλανδία σύστημα και ο ρόλος του κράτους ε, δεν είναι να αναλαμβάνει δουλειά ε, των επιχειρήσεων, αλλά να τα διευκολύνει. Ε, θα ήθελα να τονίσω επίσης και τις διασυνοριακές εργασίες και συναλλαγές, γιατί οι καταναλωτές θέλουν πλήρη εναρμόνιση, αλλά δεν έχουν και πάρα πολύ καλά επιχειρήματα Γι' αυτό δεν πρόκειται να τους υποστηρίξω σε αυτό το δρόμο. Υπάρχουν οι τροπολογίες, ε, το έχουν πει και άλλοι, ότι είναι συγκρίσιμες με άλλες τροπολογίες και υπάρχει ανάγκη ε, να γίνει καλή συνεννόηση για την αφετηρία, να ξέρουμε από πού εκινούμε. Και πολλές πολιτικές ομάδες εκφράζουν την ίδια ανησυχία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα ε, να καλυφθούν πολλές τροπολογίες από συμβιβαστικές, Οπότε τελικά να μην έχουμε 400 να ψηφίσουμε, αλλά ε, ε, είναι σε κάποιες παραδεκτές έτσι, διαστάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Good, thank you very much. Now we have... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε δύο ακόμα μιλητές. Αν όχι, θα δώσω το λόγο στην κυρία Μάινα και στον κύριο Σουβέ, ο κύριο Ζουβέ, ο κύριο Μπουδεσάρη, κάποιο άλλο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους δύο αυτούς επιπλέον ομιλητές να είναι πάρα πολύ σύντομοι, έτσι ώστε να καταλήξουν στα συμπεράσματα οι δύο εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην έκθεση του κυρίου Γκρέκα. Καταρχάς το θέμα της διαμεσολάβησης αποτέλεσε θέμα πολλών τροπολογιών. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή δεν θέλουμε να καταργήσουμε τα όσα ε, ε, υπάρχουν ε, και είναι αποδεκτά. Θα ήθελα να, να πω ότι μου φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη σχέση. Τώρα το να το κάνουμε απόλυτα υποχρεωτικό, κοιτάξτε αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσωπικά, ε, προσεκτικά γιατί η υπηρεσία πελατών μπορεί να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα σε ό,τι ε, αφορά το θέμα του κόστους ε, και εκεί υπάρχει κάποια δυσκολία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Η επιστροφή του κόστους από τον καταδικαστέντα, ένα θέμα που τέθηκε από μερικούς ε, είναι σαν να αρνείται τη φιλοσοφία αυτής της διαδικασίας που λέει ότι θα καταλήξει κανείς σε μία συμφωνία και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποιος που κερδίζει και κάποιος που χάνει. Πρότεινα μία τροπολογία σχετικά με το θέμα της, προσχώ, της πρόσβασης της ε, πληροφορίε όπου θα πρέπει ε, να είναι και ο επαγγελματία και ο εμπορευόμενο και ο καταναλωτή, όχι μόνο ο καταναλωτή, και θα ήθελα να πω δύο λόγια. Αυτά είναι ε, τροπολογίες του εισηγητή, όχι δικές μου, αλλά τι υποστηρίζω. Ε, σκέφτομαι το 92 και το 34 σε ό,τι αφορά τη σύμβαση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ενημερώνω το γίνεται περισσότερο οι καταναλωτές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι στις αποδείξεις, ε, στα τιμολόγια, παντού. Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ε, γιατί το ίδιο το σχέδιο χάνει πάρα πολύ από το ενδιαφέρον του. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπόλε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τη θαυμάσια δουλειά που έκαναν. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον κύριο Γκρέκ. Χθε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ψηφίσαμε την νομοδότηση ζώη για το ADR και επετέφθησαν συμβιβασμοί σε ό,τι αφορά σημαντικές πτυχές αυτής της οδηγίας. Ιδιαίτερα στο πεδίο εφαρμογής, στη διάρκεια, της διαδικασίας και την αντιμετώπιση των in-house διαδικασιών. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο αυτό σημείο, πετεύχθη ένα θαυμάσιο συμβιβασμό επί του άρθρου 6, το οποίο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει σχέση εξάρτησης με το νευορευόμενο υπό τον όρο που γίνονται σεβαστά ορισμένα κριτήρια τα οποία εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων η συμμετοχή σε ένα συλλογικό όργανο ή μία ε, ε, ρύθμιση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και το, ε, η επαγόρευση να λαμβάνει απευθεία εντολές και οδηγίες από τον επαγγελματία. Πρόκειται συνεπώς για ένα συμβιβασμό ο οποίος αντιστοιχεί στο στόχο εξασφάλισης ακαιρεότητας και ανεξαρτησίας των φορέων αυτών. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια λύση που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία σε αντίθεση με την άποψη που υποστηρίζει ο εισηγητής και τη στηρίζει και η Επιτροπή βάσει της οποίας η ανεξαρτησία των οργανισμών ε, ε, μπορεί να, μπορούμε να εγγυηθούμε από την αποκλεισμό από τις διαδικασίες όπου υπάρχουν διαδικασίες σύνδεσης μεταξύ αυτού που αποφασίζει και τον ενδιαφερόμενο. Από την άλλη πλευρά, αρκετές φορές επαναλάβαμε ότι και στη χώρα μου και όχι μόνο υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει μία διαδικασία συμφιλίωσης που προβλέπει μία ίση εκπροσώπηση και των δύο στα πλαίσια ενός συλλογικού οργάνου. Και αυτό εξασφαλίζει μία ισότητα στην εκπροσώπηση και των δύο μερών. Συνεπώς ε, δείχνουμε ότι η ανεξαρτησία των οργανισμών αυτών των φορέων αυτών θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μέσω ενός συλλογικού συστήματος ή μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων κριτηρίων. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια λύση σε αυτό το θέμα, γιατί θα ήταν εντελώς αρνητικό με ένα κανονισμό που θα πρέπει να διευκολύνει την ε, εναλλακτική επίλυση ε, καταναλωτικών διαφορών, ε, να δημιουργήσουμε προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά λύσεις που ήδη ε, εφαρμόζονται και που εφαρμόζονται και επιτυχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι το επεξεργάζεστε αυτό το θέμα εξ ονόματος Επιτροπής Νομοθετικών Υποθέσεων. Είστε λοιπόν ευπρόσδοκτος σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την, ε, που πήρατε το λόγο. Θα ήθελα τώρα να καλέσω την Επιτροπή να ε, πάρει το λόγο και η κυρία Μάνα και η κυρία Ρούσο. Η κυρία Μάνα, ως υπεύθυνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος Επιτροπής και η Χριστίνα θα με διορθώσει αν χρειαστεί. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, τους Σκιώδης και το προσωπικό για την εργασία τους, αλλά δεν το κάνω τυπικά. Θα ήθελα να πω ότι αυτό ε, δείχνει πόσο αυτή η εργασία, δείχνει πόσο δεσμεύονται οι μεν και οι δε και πραγματικά ασχολήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσπαθήσαμε και εμείς να τους δώσουμε τις πληροφορίες όταν χρειάζονταν τη συνεργασία μας. Για μας είναι πολύ ενθαρρυντική η σημερινή συζήτηση, γιατί φαίνουμε, φαίνεται ότι, από τη συζήτηση ότι δεν υπάρχουν ε, ουσιώδη προβλήματα και διαφορές μεταξύ μας και υπάρχει σύγκληση απόψεων σε όλο το πολιτικό φάσμα της Επιτροπής σας με, τη, με βάση τις θέσεις που εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήταν ιδιαίτερα λυπηρό να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στα πλαίσια των ε, εργασιών του σώματος. Θα θυμόσαστε ότι είναι μία από τις 12 προτάσεις της πράξης της ενίας αγοράς για γρήγορη έγκριση, όπως εκφράστηκε και σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και στο Κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής του ΕΛΚ το Φεβρουάριο μίλησε στο Κοινοβούλιο και ζήτησε τάχιστη έγκριση αυτών των προτάσεων που καταγράφονται στην πράξη ενίας αγοράς. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή σας να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και να ψηφίσετε τις δύο εκθέσεις πριν από το καλοκαίρι. Εν είδη εισήγησης, θα ήθελα να υπογραμμίσω την αρχή της επικουρικότητας. Πολύ από όσους έλαβαν το λόγο, σκιώδεις, εισηγητές και ούτω καθεξής, ε, επανήλθαν στο θέμα της επικουρικότητας. Το είχαμε κατά νου όταν συντάξαμε αυτές τις προτάσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαφορετικότητα του ADR. Δεν υπάρχουν πρότυπα Εναλλακτική επίλυση διαφορών και ούτε θέλουμε να τα επιβάλλουμε. Εμείς κρατάμε όλα τα καλά στοιχεία του ADR στα κράτη-μέλη και συμπεριλαμβάνουμε διαφορετικές προσεγγίσεις από τη διαμεσολάβηση, την ε, ανεξαρτησία, πάνελ τρίτων μερών και διαδικασία συμφιλίωσης όπως υπάρχει και υπάρχει ιδιαίτερα στην Ιταλία σε περίπτωση επίλυσης διαφόρων. Ο κύριος Βαλτασάρη συμμετείχε ενεργά και πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση λαμβάνει υπόψη την Ιταλική ιδιαιτερότητα. Ως προς το ADR, την εναλλακτική επίλυση διαφόρων. Εν συντομία, δεχόμαστε τα περισσότερα σημεία της έκθεσης ΚΡΕΚ ως προς το πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να επεκτείνουμε το ADR για να καλύπτει τις διασυνοριακές διαφορές. Εκεί που υπάρχει, που προϋπάρχει θα πρέπει να διατηρηθεί. Η διασυνοριακή διάσταση είναι σημαντική. Δεν θέλουμε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Μάλλον, για να το πω αλλιώς, ο περιορισμός του ADR θα ήταν παλινοδία. Θα οδηγούσε σε περαιτέρω κατακερματισμό και θα ε, δυναμίτιζε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ο καταναλωτής θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε επιφυλακτικοί ως προς εξαιρέσεις. Επίσης, δεν θέλουμε τομεακούς αποκλισμούς. Αλλά μπορούμε να δεχτούμε διάζουσες καταστάσεις. φύγει το ζήτημα των δέκο. Θεωρούμε ότι αποκλείονται από την οδηγία, γιατί μιλάμε για, για θέματα συμβατικής ευθύνης και συμβατικών υποχρεώσεων. Συνεπώς δεν έχουμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια των δέκο μεταξύ ενό εμπόρου και καταναλωτή, άρα δεν εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής, αλλά αν θέλετε μπορούμε να το ε, διευκρινίσουμε στην αιτιολογική σκέψη. Ως προς το θέμα των διαμεσολαβητών επιχειρήσεων, που είναι ένα γαλλικό φαινόμενο, αν και μπορεί να υπάρχουν και αλλού στην Ευρώπη, η αρχική μας πρόταση δεν περιλαμβάνει τους διαμεσολαβητές στο πεδίο εφαρμογής του ADR. Κατανοούμε τις ανησυχίες που υπάρχουν ως προσέλιψη ανεξαρτησίας, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, αλλά από ό,τι φαίνεται η επικουρικότητα λειτουργήσε καλώς σε σχέση με συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών και θα πρέπει να υπάρχουν σωστές διασφαλίσεις που να εντάσσονται στο κείμενο. Ως προς την υποχρέωση του καταναλωτή να επανέλθει στον έμπορο πριν εκινήσει τη διαδικασία ADR, για μας είναι ένα θέμα επικουρικότητας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε έναν κανόνα στην οδηγία που, που ίσως τρευλώσει τα ε, πρότυπα ADR, τα σχήματα ADR που λειτουργούν σωστά. Επειδή συμφωνούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το πρώτο βήμα είναι να ε, αποτανθεί κανείς στον έμπορο, ο καταναλωτής δηλαδή στον έμπορο, γιατί αυτό είναι υπέρ του καταναλωτή, είναι ο γρηγορότερος τρόπος επίλυσης. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, αλλά αν θέλετε θα το εντάξουμε στην αιτιολογική σκέψη. Στο άρθρο 5 υπάρχουν οι κατάλληλες, οι σχετικές διατάξεις ως προς τη διαδικασία. Εάν ένας οργανισμός ADR έχει μια τέτοια υποχρέωση, τότε παραμένει. Αλλά δεν θα θέλαμε να υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για όλα τα εναλλακτικά σχήματα επίλυσης διαφορών. Αν υπάρχει στα κράτη-μέλη, ας παραμείνει. Ως προς τις πληροφορίες, ο κύριος Ζουβά πολύ σωστά παρενέβη και είπε ότι η πληροφόρηση του καταναλωτή είναι ουσιώδες τμήμα αυτής της πρότασης. Θέλουμε ο καταναλωτής να έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το εύκολο και απλό μέσο φιλικό προς τον καταναλωτή, μέσο επίλυσης διαφοράς. Δηλαδή θα μπορεί όταν αποτανθεί στον έμπορο να του πει λύστε μου το πρόβλημα, διαφορετικά θα προσφύγω στο επόμενο μέσο που έχω στη διάθεσή μου. Ε, δεν θα ε, προσφύγω στη δικαιοσύνη, άρα ε, δεν θα υποβληθώ σε έξοδα. Υπάρχει ένα πολύ πιο απλό μέσο που είναι το ADR. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ καλά πληροφορημένος ο καταναλωτής. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενταχθεί στην οδηγία και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει διοικητικός φόρτος ή θα επιβάλλει διοικητικό φόρτο στους εμπόρους. Ως προς τις δαπάνες επανέρχομαι στην επικουρικότητα. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας στα κράτη-μέλη. Ε, πολλές φορές δεν υφίσταται κόστος, υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση των εθνικών ATR ανάλογα με τα κράτη και ανάλογα με τον τομέα. Άρα θέλουμε να είναι ολιγοδάπανη η διαδικασία ή καθόλου δαπανηρή και εν πάση περιπτώσει αυτό εμπίπτει στα εθνικά πλαίσια ως προς την αρχή του ότι αυτός που χάνει την υπόθεση καταβάλει τα έξοδα Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία αφορά ένα δικαστικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι όμως ένα δικαστικό πλαίσιο επίλυσης. Δεν πρόκειται για ένα εθνικό δικαιοδοτικό σύστημα. Δεν είναι κάτι τέτοιο το ADR. Είναι διαφορετική προσέγγιση, έχει διαφορετικό DNA αν θέλετε να σας το πω και έτσι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε ποιος έχει κερδίσει την υπόθεση και ποιος την έχει χάσει ως προς την ανεξαρτησία, αμεροληψία, νομιμότητα και ελευθερία. Εδώ υπάρχει συνένεση. Τώρα, να στραφούμε στις ηλεκτρονικές επιλύσεις, στην έκθεση των. Υποστηρίζουμε τη θέση της εισηγήτητας, της εισηγήτητας ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, απλούστευση και σαφήνεια στις επιλύσεις. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για απλούστευση, έτσι ώστε το κείμενο να είναι ευνόητο και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, μιλάμε για σημεία σύνδεση, σημεία επαφής, ε, ε, ε, διαμεσολαβητές. Ίσως έχουμε επιμείνει υπερβολικά σε αυτά, και μπορούμε ε, ίσως να μιλήσουμε για πολλαπλούς παίχτες ε, έτσι ώστε το όλο πλαίσιο να είναι ευνόητο για τον καταναλωτή. Ως προς τη μετάφραση θα πρέπει το πλαίσιο να είναι φιλικό προς το χρήστη, άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να κατανοεί ε, εύκολα το όλο πλαίσιο να είναι εύχριστο και ούτω καθεξής. Στις συζητήσεις με την εισηγήτρια τις ε, δώσαμε εγγύηση σε σχέση με τα μηχανήματα μετάφρασης, αλλά τα μηχανήματα έχουν και όρια και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο το οποίο να μπορεί να χειριστεί όχι μόνο τις παρεξηγήσεις που σχετίζονται με την χρήση διαφορετικής γλώσσας, αλλά και τις πολιτισμικές διαφορές που εγείρονται μεταξύ ενός καταναλωτή σε μία χώρα και ενός έμπορου σε μία άλλη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής, ο οποίος να μπορέσει να βοηθήσει στην επίλυση της διαφοράς. Διαφωνούμε με την εισηγήτρια σε ένα σημείο. Η πλατφόρμα ODR δεν θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω της δικτυακής πύλης Europe. Το συζητήσαμε στην Κομισιόν και θεωρούμε ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος χειρισμού Το Yuri Europe είναι μία πύλη πληροφόρησης και χρειάζονται αρκετά κλικαρίσματα έτσι ώστε να φτάσετε στην πλατφόρμα. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε το Solvit που έχει αρκετά links και μπορείτε να φτάσετε σε αυτό και από το Yuri Europe αλλά και με διαφορετικούς τρόπους και άμεσα από τις δικτυακές πύλες του εμπόρου. Δηλαδή μπορείτε να το κλικάρετε από την πύλη του εμπόρου. Ως προς τις προθεσμίες, οι 30 ημέρες είναι μια φιλόδοξη προθεσμία, αρκετά φιλόδοξη, αλλά μπορούμε να σταθούμε ευέλικτοι και ως προς την ανάγκη προστασίας προσωπικών δεδομένων θεωρούμε ότι είναι ύψης της σημασίας, φυσικά και συμφωνούμε και είμαστε σε επαφή με την Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Επιτροπή. Ελπίζω να σας απάντησα. Σας ευχαριστώ. Καλύψατε πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήσατε το θέμα. Και έχει πάει τα ώρα περίπου. Θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας για να ολοκληρώσουν οι κυριατούν και μετά ε, ο άλλος εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους. Ας επικεντρωθούμε σε ορισμένα θέματα καταναλωτής, επιχείρηση, επιχείρηση, καταναλωτής. Εάν ορισμένες ADR έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε επίλυση των διαφορών με την παρέμβαση, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τους αποκλείσουμε για να μην ε, καταστρέψουμε αυτή την προστιθέμενη αξία που υπάρχει σε πολλές χώρες. Συνεπώς ε, ας διατηρήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό αν αυτά τα Τα NDR ε, είναι λειτουργικά. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στη λέξη διαμεσολαβητής. σύμβουλοι θα έλεγα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το διαμεσολαβητής. Στην ουσία είναι σύμβουλοι. Σε ό,τι αφορά την ε, παρατήρηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί, έχει ληφθεί υπόψη αυτό το αίτημα στην τελευταία αυτή έκθεση. Έγινε αναφορά στο διάστημα των 30 ημερών. Θα πρέπει όμως να συγχρονίσουμε και το χρόνο που προβλέπετε για τον οργανισμό EDR. Συμπεριέλαβα τα ίδια προαπαιτούμενα και στην έκθεση για το ADR. Τελευταίο σημείο, την προσβασιμότητα, έτσι την ονομάζουμε, accessibility. Μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης, του πόρταλ, μιλάμε πάντοτε για μια ελεύθερη, για μια εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες. Ενδεχομένως εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Αυτή η πληροφορία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από παντού. Δεν είναι το θέμα μόνο να χρησιμοποιήσει κανείς το ευρωπαϊκό σύστημα. Υπάρχουν διάφορα links τα οποία θα μπορούσαν να είναι παντού. Αν βρισκόμαστε στη σελίδα Euro Europe, Εκεί μπορούμε να βρούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, πληροφορίες για το ADR και διάφορα άλλα. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο ADR, εάν παράλληλα υπάρχει και ε, ε, ο μη ηλεκτρονικός φορέας ε, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορεί να δουν ότι υπάρχει μία πληρή και χρησιμοποιούν είτε την, τον ηλεκτρονικό είτε τον ελλακτικό φορέα. Δεν θα ήθελα να προσθέσω άλλα ε, ε, δεν θα ήθελα να υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, θα ήθελα να υπάρχει ένα σημείο εύκολης πρόσβασης που μας επιτρέπει να ε, βρούμε άμεσα τις πληροφορίες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι μια αναγκαία λύση. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά θέματα χρόνου και εγώ είμαι υπέρ του να κινηθούμε ταχαίως. Σε ό,τι αφορά την ε, αυτόματη μετάφραση, δεν υπάρχει μια ήδη έτοιμη λύση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα επιταχύνουμε τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση αφήνω αυτό το σημείο για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Λουί Γκρέκ. Νομίζω ότι θα είμαι πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο χρόνο πιέζει. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε, όχι να κατασκευάσουμε, να καταστρέψουμε αυτά που ήδη είναι λειτουργικά. Σε γενικές γραμμές θα ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ σε ό,τι αφορά διάφορα θέματα, το in-house mediation, τη διαμεσολάβηση από την επιχείρηση. Το δεύτερο σημαντικό σημείο που αναφέρθηκε αφορούσε τη συνδιαλλαγή και όχι την αντιπαράθεση. Νομίζω ότι αν το ξεχάσουμε αυτό, ξεχνάμε την όλη διάσταση του θέματος στους τομείς, όπου είναι, το, θέμα είναι γλωσσικό. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε τη σωστή διατύπωση, τη σωστή μετάφραση και να επιτύχουμε μια συμφωνία με, ε, με τους περισσότερους. Σε ό,τι αφορά το θέμα άλλων αρχών, άλλων θεμάτων, η πληροφορία. Η πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική σε τομείς όπου πιστεύω ότι αναφέρθηκαν πολλά σε ότι αφορά την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου. Νομίζω ότι αυτό το αναφέραμε ήδη στα εκτιμώντας, το αναφέραμε ήδη στο άρθρο και νομίζω ότι σαφώς είναι σαφείς οι προθέσεις μας. Δεν θέλουμε όμως να είναι υποχρεωτικό για τον καταναλωτή να επικοινωνήσει προηγουμένως με τον έμπορο. Σε γενικές γραμμές κύριε Πρόεδρε δεν νομίζω ότι υπάρχουν μείζονες διαφορές. Παρόλα αυτά, εάν οι συνάδελφοι, αν οι σκιώδεις συζητητές θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επίτευξη ενός καλύτερου συμβιβασμού που ε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη νομοθετική πρόταση, θα είμαστε έτοιμοι να το λάβουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Χαίρομαι που μπόρεσε να τελειώσει η συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του διερμηνείς που μένουν λίγο παραπάνω. Η πρότασή μα είναι να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση στις 9 Ιουλίου για τι ε, τροπολογίε ε, συμβιβασμού. Οι συγκητές ε, και σκιώδει συγκητές θα συναντηθούν. Από πλευρά μου πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει όμω να δείτε πώς, τι θα γίνει με του συμβιβασμού. Έχουμε όμως ε, προβλέπεται αυτό ο επιπλέον χρόνος για να μπορέσετε να το συζητήσετε πριν την ψηφοφορία που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Βεβαίω, αν θα θέλετε να κάνετε αλλαγέ, θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μάινα, την κυρία Ρούσο. Το επόμενο θέμα, έκθεση του κυρίου Ροσφόρ για τα προγράμματα των καταναλωτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα ξαναδούμε την κυρία Μάνα ή κάποιον άλλον από την ομάδα της ε, σε κάθε περίπτωση. Περιμένω να τα ξαναπούμε στις 3. Ευχαριστώ πολύ.